No hammer today? No hammer? Fine. You have to switch on the other. Yes. Yes. This is going to be the one. Buenos días. Καλημέρα σας. Να σας καλημερίσω. Muy buenos días, queridos colegas. συνάδελφοι. Κυρίε και κύριοι, επειδή δεν έχω το σφυρί εδώ στο Προεδρείο για να επίστησω την προσοχή σας, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε να μας βοηθήσετε για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω το εξή. Όλοι όσοι δεν ήσασταν παρόντες στην καταστατική συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για αυτό το δεύτερο ημις της μας, θα ήθελα εκ μέρους μου προσωπικά και εκ μέρους όλων των μελών του Προεδρείου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την επανεκλογή μας ώστε να προεδρεύσουμε και για το δεύτερο ήμιση της θητείας ε, της Επιτροπής μας. Θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε διδάγματα από την εμπειρία που αποκομίσαμε ως τώρα. Αυτό τι σημαίνει πρώτα απ' όλα. Να τηρούμε τους χρόνους. Έχουμε μια πολύ βεβαρημένη σε διάταξη με 25 σημεία. Όχι, λίγα λοιπόν. 25 σημεία. Σας παρακαλώ λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εμείνουμε στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για το κάθε σημείο για να ολοκληρώσουμε. Τούτων λεχθέντων, να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπότσκοφ, τον ε, Υπουργό Δικαιοσύνη της Δανίας, εκπροσωπεί την ε, Δανική Προεδρία του Συμβουλίου. Να τον καλωσορίσουμε, είναι τιμή και χαρά για μας να σας έχουμε μαζί μας και βεβαίως να πω ευθύς εξ αρχή ότι και η Επιτροπή Λίμπια στο σύνολό αλλά και κάθε μέλος χωριστά θέλουμε να σα προσφέρουμε κάθε δυνατή συνεργασία ώστε να στεφθεί με επιτυχία η Προεδρία σα. Πριν δώσουμε το λόγο να κάνει την παρουσίαση στον κύριο Μπότσκοφ, θεωρώ δεδομένο ότι υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη. Το σημείο υπαριθμών 20 για τη Συμφωνία της Ένωσης με τον Καναδά για τη μεταφορά των δεδομένων PNR που προβλέπεται σήμερα στηθεί από τις 17.45 έως 18.30 θα γίνει και κλεισμό των θυρών. τη η σε διάταξη και κρίνουμε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων που βλέπετε στον κατάλογο των πέντε αυτών συνεδριάσεων. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνουμε αυτά τα πρακτικά. Υιοθετούνται λοιπόν και να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Μπότσκοφ, τον Δανό Υπουργό Δικαιοσύνη, να μας παρουσιάσει τα θέματα προτεραιότητας της Δανικής Προεδρίας για το εξάμεινο αυτό. Μετά από την παρουσίαση του Υπουργού θα δώσω το λόγο για ερωτήσεις και μετά θα απαντήσει ο υπουργό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Chairman, and uh, once Πρόεδρε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την επανεκλογή σας θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής. Προσβλέπω σε μια πολύ καλή συνεργασία με ολόκληρη την Επιτροπή φυσικά. Τώρα μου επιτρέπετε θα μιλήσω τη γλώσσα μου για να κάνω την παρουσίασή μου. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας μας σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα. Μεγάλη τιμή λοιπόν για μένα. Αναλαμβάνω λοιπόν την Προεδρία με πολλά θέματα μπροστά μου. Θα σα διαβεβαιώ ότι θα την κάνω στον βέλσο των δυνατοτήτων μου. Έχω ήδη κάνει επαφέ με κάποιου από εσάς ε, και στις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο έχουμε συναντηθεί σε πολύ καλές επικοδομητικέ συνεδριάσεις ε, οι οποίες μας επέτρεψαν και αμοιβαία συνεννόηση και έναν ειλικρινή διάλογο. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε σε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, σε πολύ καλό κλίμα του επόμενου μήνε. Ω πρόεδρος λοιπόν θα ήθελα να ως Προεδρεύων θα ήθελα πάνω απ' όλα να εντατικοποιήσω τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όσον αφορά τις δράσει που θα αναλάβουμε, θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι έχουμε αποφασίσει να βελτιστοποιήσουμε τη συνεργασία και με δικαστές και άνθρωπους ε, που έχουν ευθύνη στον τομέα αυτών, ε, μέσα από τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα των εργασιών μας. Οι άλλοι υπουργοί της Δανίας, η αντιπροσωπεία, μόνιμη αντιπροσωπεία της Δανίας, το Συμβούλιο, το προσωπικό, θα ε, εργαστούν σκληρά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Και επιτρέψτε μου να απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη της Επιτροπής σας για επαφές με μέλη του Συμβουλίου, της Προεδρίας συγκεκριμένα, εάν έχετε οποιαδήποτε επιθυμία για συζήτηση, για ενημέρωση. Το Συμβούλιο για σας έχει πάντα τις θύρες του ανοιχτέ και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. από οποιοδήποτε θέμα έχουμε στις αρμοδιότητές μας. Και επιτρέψτε μου να ε, συζητήσω τώρα, να αναφέρω τώρα κάποια από τα θέματα που θα έχουν σημασία ιδιαίτερη και θα απασχολήσουν την Προεδρία μας. Υπάρχουν και άλλα θέματα βεβαίω ε, και πολύ ευχαριστώ να τα συζητήσουμε αν θέλετε. Ω εκ τούτου, εάν ε, δείτε ότι παραλείπω κάποιο από τα θέματα που σα ενδιαφέρει, παρακαλώ ε, διατυπώστε τι ερωτήσει και τι παρατηρήσει σα. Πάντω, εγώ από πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχω τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα από την Προεδρία αυτή. Αναλαμβάνει λοιπόν την Προεδρία του Συμβουλίου η Δανία σε μια χρονική περίοδο όπου είναι ιδιαίτερα αισθητή η ανάγκη για στενή, για ουσιαστική συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ορίζει, περιγράφει ένα πλαίσιο το οποίο περικλεί ουσιαστικά κάθε τομέα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει οποιαδήποτε μας δράση να εξαρτάται από αυτό να υπάγεται σε αυτό. Φυσικά έχουμε ιδιαίτερες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε στον τομέα της ε, δικαιοσύνης και των εσωτερικών. Φερρυπίνα στην ε, μετανάστευση και το άσυλο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες θα είναι να ε, προχωρήσουμε όσο το δυνατόν προς σύναψη στην τελική του μορφή ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θα εργαστούμε σκληρά για να επιτύχουμε το στόχο αυτό εφέτος. Και θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όσο το δυνατόν περισσότερα νομοθετήματα ε, συζητήσουμε. Το Συμβούλιο έχει σημαντική πρόοδο σημειώσει ως προς την οδηγία, ε, ως προς τη συμφωνία του Δουβλίνου αλλά και την οδηγία για την υποδοχή των ετούντων και προσπαθούμε να προχωρήσουμε όχι μόνο αυτές τις, ε, αυτά τα νομοθετήματα αλλά και κάθε άλλο σχετικό νομοθέτημα. Πρέπει πάντοτε με ιδιαίτερη εστίαση των προσπαθειών μας να επιδιώκουμε συστήματα που ουσιαστικά θα προσφέρουν την προστασία σε όποιον την έχει ανάγκη. Σήμερα λοιπόν μπορώ να σας πω ότι η σημερινή μέρα έχει μια μεγάλη σημασία διότι έρχεται, τίθεται σε ισχύ σήμερα η ενισχυμένη οδηγία προς την προστασία των ε, προσφύγων. Ε, έχουμε δηλαδή ένα από τα τελικά κείμενα του συστήματος που θα συμπληρώσουν το σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιδείξει την αλληλεγγύη της με τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα, τις περισσότερες προκλήσεις, δηλαδή τις περισσότερες ροές αιτήσεων ασύλου αλλά και ε, λάθρο μεταναστών. Αυτά είναι προβλήματα κοινά, κοινά σε όλους μας. Εάν ε, το καταρρεύσει το σύστημα ασύλου της μίας χώρας, έχουμε όλοι πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει από κοινού να επιλύσουμε τα ζητήματα. Συνεργασία. Η λέξη συνεργασία δεν είναι μόνο μία λέξη, δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Συνεπάγεται συγκεκριμένες ε, δράσεις, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτά πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε διεξοδικότερα. όταν μιλάμε για διεξοδικέ δράσεις, για συγκεκριμένε δράσεις και πρωτοβουλίες, Μπορώ να σας ανακοινώσω ότι πρόκειται να γίνει μια ε, συνάντηση στην Κοπεχάγη σε μερικές ε, ημέρες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα και έχουμε και την εντολή να συζητήσω μαζί σας ε, το ε, κοινό πρόγραμμα για επανεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιστεύω θα διευκολύνει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα της ε, επανεγκατάστασης για πρώτη φορά. Εμείς στη Δανία έχουμε μακρά παράδοση βέβαια της επανεγκατάστασης. Όταν μιλάμε για μετανάστευση, μετανάστευση και ασύλο, έχουμε ήδη πολύ μεγάλη εμπειρία από διαπραγματεύσεις και με τρίτες χώρες. Επί τη βάση λοιπόν της ε, ανακοίνηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στρατηγική και τη μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να ενισχύουμε τη συνεργασία ε, με τις ε, τρίτες χώρες, ε, πράγμα το οποίο άλλωστε υπεγράμισε ως ανάγκη και η Αραβική Άνοιξη. Στο θέμα της θεώρησης διαβατηρίων έχουμε πολλά σημαντικά θέματα να ε, αντιμετωπίσουμε, όπως παραδείγματι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία επεξεργαζόμαστε για μια τροποποίηση του κανονισμού για θέματα θεώρησης διαβατηρίων, που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο την Άνοιξη. Επίσης, επεξεργαζόμαστε μία πρόταση συγκεκριμένη, εστιασμένη, αλλά και διαφορετική για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και τις σχετικές αλλαγές βέβαια που θα χρειαστούν στο σύστημα Schengen και τον τρόπο λειτουργία του. Προτεραιότητά μα είναι να ενισχυθεί η συνεργασία Schengen. Η συνεργασία Schengen έχει υποστεί σημαντικέ πιέσει τον τελευταίο καιρό. Και έτσι πρέπει να ε, συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για να βεβαιωθούμε ότι, θα πρέπει, ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία Schengen, να την αξιοποιήσουμε καλύτερα. Η συνεργασία Σέγγεν αποτελεί βάση και εγγύηση της ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων. Αποτελεί ακρογωνία ολίθο της ευρωπαϊκής μας συνεργασίας. Και μια βασική αρχή, την οποία ξέρω ότι ενστερνίζεται θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερω η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, είναι αυτή που μας οδηγεί σε προτεραιότητα στις προτάσεις εκείνες μέσα στο ε, πακέτο του Σέγγεν, ώστε να βρεθούν οι σωστές λύσεις και πάνω απ' όλα η σωστή ισορροπία, η ορθή ισορροπία μεταξύ ε, και της ανοιχτής προσέγγισης αλλά και της ε, ε ισότιμης μεταχείρισης και της ασφάλειας. Αυτές είναι οι προσπάθειες που θα ε, μας απασχολήσουν ε, και η ασφάλεια βεβαίως, η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, η αστυνομία, το ποινικό δίκαιο, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με τα προβλήματα της ε, τρομοκρατίας και της υπερσυνοριακής εγκληματικότητας. Δυστυχώς ακόμη αυτή αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς ως πολιτικοί υπεύθυνοι είμαστε υποχρεωμένοι να, να συνεργαστούμε, να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε την, την ε, απειλή αυτή και να ε, επιτελέσουμε σε τελευταία ανάλυση το έργο το οποίο απαιτεί ο πολίτη κατά τρόπο επιτυχή. Για να είμαστε όμω επιτυχεί στον τομέα αυτό, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι συνεργαζόμαστε στενά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε στενή συνεργασία να εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες ε, συνθήκες ε, συνεργασίας πέραν των συνόρων ε, με τα κατάλληλα μέσα μεταξύ των αρχών μας. Και έτσι προτείνουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει με την ε, συνεργασία αυτή να καταπολεμήσουμε και τη δημοκρατία και την ε, διακίνηση ανθρώπων, του εμπόριου ανθρώπων. Ελπίζουμε να θα εξασφαλίσουμε γρήγορα πρόοδο στα θέματα αυτά με ορθή ισορροπία, με κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής εφαρμογής νομοθεσίας και ταυτόχρονα της προστασίας των βασικών αρχών του ιδιωτικού βίου. Οι ρυθμίσεις που θα εισαχθούν θα πρέπει να περιοριστούν στο απολύτως απαραίτητο για την επιτρέψη του αποτελέσματος. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να αποτελέσει ε, λευκό επιταγή για την εισαγωγή ε, περιοριστικών ε, διατάξεων. Αλλά πάλι θέλουμε να είμαστε και πολύ αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση τρομοκρατία και του υπερσυναριακού εγκλήματος. Μιλάμε λοιπόν για την πρόταση αυτή, την πρόταση PNR, η οποία δεν θα πρέπει να ε, οδηγεί σε ευρωπορίες πέραν του απολύτω απαραίτητου στη διάθεση των πληροφοριών από τη μια αρχή στην άλλη και από την άλλη κάθε τύπου πληροφορία την οποία δεν απαιτείται να γνωρίζει ε, η αρχή, η υπεύθυνη αρχή, η αστυνομική αρχή δεν θα πρέπει να συλλέγεται. Αυτή είναι η βασική αρχή που ακολουθούμε. Πιστεύω ότι ε, μας εξασφαλίζει τη χρυσή τομή, την, ε, τη λεπτή αυτή ισορροπία και πιστεύω ότι μπορούμε να καταθέσουμε συγκεκριμένε προτάσεις στην υπόθεση αυτή. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε τώρα, να στραφώ σε ένα άλλο σημαντικό θέμα για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, PNR, με την συμφωνία τη σχετική με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουμε συνάψει για ανταλλαγή πληροφοριών και η οποία ε, θα έρθει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες. Θα θέλω να επισημάνω ότι σε διαπραγματεύσεις ε, διεθνείς δεν είναι δυνατόν κανείς να περιμένει ότι θα εξασφαλίσει ε, κάθε του διεκδίκηση μέσα στη τελική συμφωνία. Αυτό λοιπόν ισχύει και στις ε, διαπραγματεύσεις μας με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, πιστεύω ότι το σχέδιο συμφωνίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, το πρώτο σχέδιο συμφωνίας, είναι το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε σχέση με το όσο θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε αυτή την εποχή, αυτό τον καιρό. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι βελτιώσεις που επετεύχθησαν στο κείμενο της συμφωνίας σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην αιμονή και την επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Του τουλεχθέντος πιστεύουμε και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την σύναψη αυτή της συμφωνίας. Η ΔΕ Προεδρία από πλευρά της είναι στη διάθεσή σα για να συζητήσει εάν μπορούμε να προσφέρουμε είτε εμείς είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις του σημαντικού θέματος. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα εγείρουμε είναι το θέμα των πρόδρομων ουσιών για εκρηκτικά. Το θέμα των εκρηκτικών είναι, οι πρόδρομε ουσίε μάλλον εκρηκτικών, είναι ένα από τα μέσα που προτιμούν ιδιαίτερω οι τρομοκράτε ε, για τι δημοκρατικέ του επιθέσει. Ω εκ τούτου, οι πρόδρομε αυτέ ουσίε που έχουν και αντικείμενο συζήτηση για αρκετό καιρό πρέπει πλέον με υπευθυνότητα να αντιμετωπιστούν, να εγκριθεί δηλαδή το σχετικό ευρωπαϊκό νομοθέτημα. Η δε καλύτερη μέθοδος ώστε να αποφευχθεί η εγκληματικότητα επισημένο είναι πάνω απ' όλα όχι η καταστολή αλλά η πρόληψη. Αυτό ισχύει και για την τρομοκρατία βεβαίως. και για τις ε, άλλες εγκληματικές δραστηριότητες του κοινού ποινικού δικαίου. Έτσι λοιπόν, επικεντρωνόμαστε στον καλύτερο, στους καλύτερους δυνατούς τρόπους αφενός να αποτρέψουμε τη στροφή προς την ακρότητα, την ακέραιοφροσύνη των νέων μας, αφετέρου δε να ε, επαναφέρουμε στον ορθό δρόμο όσους νέους έχουν ενδεχομένως βρει αυτόν τον δρόμο της ακεραιοφροσύνης, της ακρότητας δηλαδή. Σε αυτό στηριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό και στην ε, απόφαση ε, τη δικαστική απόφαση για την ε, διεξαγωγή ανακρίσεων, προανακρίσεως, που θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες των ε, διοκτικών μας αρχών στη διερεύνηση εγκλημάτων, όχι με νέα μέσα, αλλά με πιο αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων μέσων. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να στραφούμε και προς την κατάσταση του θύματος μια εγκληματική δραστηριότητα. Άρα θα δώσουμε όθηση και σε μια δέσμη μέτρων που αφορούν τα θύματα, είτε σε αυτόν τον τομέα είτε σε άλλου. Η πρόκληση που αντιμετωπίσουμε είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, αλλά και ταυτόχρονα να ε, μην παραβιάσουμε, να εξασφαλίσουμε την απόλαυση από τον ε, κατηγορούμενο των δικών του δικαιωμάτων, να μην παραβιαστούν δηλαδή τα δικά του δικαιώματα. Και πάντοτε με όλες τις ε, καλύτερες προθέσεις του κόσμου δεν θα, δεν πρέπει και να παραγνωρίζουμε την, το, το νομικό πλαίσιο μας στο οποίο κινούμαστε, την πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στην νομοθεσία για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και τη σχετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου που επανέρχεται στο Συμβούλιο τώρα. Ε, προβλέπεται ότι θα είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσει, σκληρέ οι διαπραγματεύσει. Σε άτυπο επίπεδο ε, διαρευνούμε το πεδίο, βολιδοσκοπούμε του συναδέλφου. Η, Ευρω... η Δανική Προεδρία σκοπεύει να δώσει μεγάλη μάχη στην υπόθεση αυτή με όλε τι δυνάμει. Και ξέρω βέβαια ότι είμαστε πολύ φιλόδοξοι, αλλά φιλόδοξους στόχους έχουμε διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικά τα ζητήματα που ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και πιστεύουμε επίσης ότι αν συνεργαστούμε όλοι καλά μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι η Προεδρία της Δανίας στο Συμβούλιο μπορεί να μπορεί να αποτελέσει μάλλον ε, ένα νέο σταθμό για καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον, με, ανοιχτή, ε, με ανοιχτό διάλογο, με καλή συνεργασία σε κάθε επίπεδο, με συνεργασία που θα φέρνει αποτελέσματα, αυτό επιδιώκουμε, και αυτό σημαίνει καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αναλάβει αποφάσεις σημαντικές. Είναι υποχρεωμένη να λάβει αποφάσεις σημαντικές για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας μας. Και πιστεύω ότι εμείς μαζί μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που θα αλλάξει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ είμαι ε, ακριφνής υποστηριχτής του ιδεώδους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω όμως ότι πέραν αυτού και πέραν των ιδεωδών θα πρέπει να κρυθούμε με βάση τα όσα έχουμε επιτύχει, με βάση τα όσα κάνουμε στην πράξη. Ας ανασκουμποθούμε λοιπόν, ας ε, συνενωθούμε, ας συνεργαστούμε και ας αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις. We thank you. We thank you. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Δανέζικης Προεδρίας του εξαμένου αυτού. Και τώρα ας ξεκινήσουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα έλεγα ο καθένας δύο-τρία λεφτά να μιλήσει, ο κάθε δηλαδή συντονιστής, κάθε εκπρόσωπος των πολιτικών ομάδων και μετά θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων, αφού πρώτα μας απαντήσει ο υπουργό για τους ευρωβουλευτές. Μην ξεχνάτε την πίεση του χρόνου. Σας είπα από την αρχή ότι πιεζόμαστε από τα 25 σημεία της ημερήσιας διάταξης. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα διεκπαιρεώσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι μετά έχουμε και τη συνάντηση των συντονιστών σήμερα το πρωί. Ο κύριος Μπουσουτήλ από το ΕΛΚΑ είναι ο πρώτος συντονιστής. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Εκ μέρους του ΕΛΚΑ θα ήθελα να σας απευθύνω α, τις διαβεβαιώσεις για στενή συνεργασία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας ήδη ξεκίνησε καλά. Βρήκατε το χρόνο να συναντήσετε τους συντονιστές ατομικά, τον καθένα. Συναντηθήκαμε χθε και νομίζω ότι είναι ένα θαυμάσιο τρόπος για να ξεκινήσει η συνεργασία μας. Ε, ίσως καλό θα ήταν, ε, αν μπορούσα να σας ε, πείσω, να ξεφορτωθείτε το out ε, στον τομέα της δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων, εσείς ως Δανία εννοώ. Να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΕΛΚΑ. Ελπίζουμε η Προεδρία σας θα μας βοηθήσει από τους τομείς. Καταρχάς, στον τομέα της κοινή πολιτικής ασύλου. Ξέρετε ότι φέτος, ε, το 2012, είναι ο στόχος μας για να πετύχουμε μια τέτοια πολιτική, πραγματική πολιτική, ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Ξέρετε επίσης ότι αυτή η πολιτική έχει κολλήσει. Υπάρχουν βαθιές διαφορές ανάμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών και στο Κοινοβούλιο για την ουσία που θα πρέπει να διαπνέει αυτή την κοινή πολιτική. Δηλαδή, πώς ε, οι χώρες μπορούν να δρουν από κοινού ε, εκφράζοντας πλήρη αλληλεγγύη η μία προς την άλλη σε αυτόν τον τομέα. Πέστε μας, τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα πάρει η Δανέζικη πρωτοβουλία στον τομέα της πολιτικής ασύλου για να απεμπλέξει αυτό το αδιέξοδο και να εκφραστεί πραγματική αλληλεγγύη. Κάτι άλλο σημαντικό για μας είναι το Σέγγεν βέβαια. Και καλωσορίζουμε την αλλαγή πολιτικής που έχει παρουσιάσει η κυβέρνησή σας σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς ε, που είχαμε, που είχαμε δει από τη Δανία στη ζώνη Σέγγεν. Και ελπίζουμε η Προεδρία σας να βοηθήσει ούτως ώστε να ενισχυθεί η περιοχή του Σέγγεν και να μην δεχθεί πιέσεις και επιθέσεις. Ένα άλλος τομέας που μπορεί να σημειωθεί πρόοδος είναι ε, η Ευρωπαϊκή Εντολή Ανακρίσεων. Έχουμε μια έκθεση η οποία μόλις παρουσιάστηκε από τον συνάδελφο τον κύριο Μέλο και ελπίζουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό με βάση αυτή την έκθεση, κοινοβούλιο και συμβούλιο δηλαδή, και βεβαίω το πακέτο για τα θύματα, στο οποίο εσείς αναφερθήκατε. Τέλος, ελπίζουμε ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος και στη συμφωνία για το PNR, για το Passenger Name Record και θα υποστηρίξουμε την ανάγκη για στενή συνεργασία με άλλες χώρες και μεταξύ βεβαίως των κρατών μελών ε, στον ε, αυτόν τον αγώνα καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας αλλά με βάση μην ξεχνάμε όμως και τα και τις αρχές που είναι πολύ σημαντικές για μας, ε, το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Μωράης. Ευχαριστώ κύριε Μπότσκοφ. Από τους σοσιαλιστές. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις ε, συναντήσεις που είχαμε το 2011 και για τη χθεσινή συνάντηση. θα επαναλάβω κάτι που είπαν όλοι οι συντονιστές αυτή τη συνάντηση που είχατε και που δείχνει ότι Υπάρχουν ένα-δύο θέματα. εσεί και η Δανέζικη Προεδρία προσπαθείτε να καλύψετε όλο τον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων ε, του επόμενου έξι μήνε, τη δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά έχουμε μάθει ότι μέσα σε μια εξάμεινη προεδρία κανεί δεν μπορεί να τα πετύχει όλα και πρέπει να βάλετε κάποιε προτεραιότητε, ώστε εκεί να σημειωθεί πρόοδο. Οι τομεί όπου υπάρχει μια κάποια απογοήτευση σε όλους ε, είναι καταρχάς ο τομέας, το πακέτο του ασύλου, είναι προτεραιότητα όχι μόνο για τους σοσιαλιστές, αλλά για όλες τις πολιτικές ομάδες και εκεί υπάρχει κόντρα με το Συμβούλιο. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις, ε, πολλές αναδιατυπώσεις. Ξέρετε πολύ καλά την ιστορία του πακέτου ασύλου και ζητάμε από την Προεδρία σας τουλάχιστον να σημειωθεί α, πρόοδος ε, στο θέμα αυτό του και το συζητήσαμε στις δύο προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε. Πάντως, ε, δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, είναι προτεραιότητα για μας. Για το θέμα του Σέγγεν, επίσης. Η Δανία έχει εμπλακεί πολύ στο θέμα του Σέγγεν. Τα βασικά θέματα για μας δεν είναι μόνο απλώς να σημειωθεί η πρόοδος, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Καταλαβαίνουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να εξασφαλίσουν εσωτερική τους ασφάλεια, αλλά όπως μας εξήγησαν και οι Δανείοι τους τελευταίους ε, ε, μήνες, ε, θα πρέπει να υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και εμπλοκή και αυτό σημαίνει εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Για την πρόσβαση στα δεδομένα και το θέμα της διαφάνειας. Η Δανία έχει απίστευτο ιστορικό στα θέματα της διαφάνειας ε, εσωτερικά. Και νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξει το θέμα της πλειοψηφίας των δύο τρίτων, με την οποία το Κοινοβούλιο ε, το Δεκέμβριο υιοθέτησε αυτή την θέση στην έκθεση Κάσμαν. Θέλουμε να το σπρώξουμε και να περάσει από το Συμβούλιο. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τη διαφάνεια στα διάφορα κράτη-μέλη, το ξέρουμε αυτό, αλλά η Δανία τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Είναι οι δήμονες και επομένως θέλουμε να το, να σπρώξετε αυτό το θέμα, να το περάσετε από το Συμβούλιο. Ε, ένα θέμα που δεν έφερε ο κ. Μπουσούτηλ, ο προηγούμενος ομιλητής, ε, και που είναι δύσκολο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στα εν μέσω και σοβούσεις της ε, οικονομικής κρίσης, είναι η νόμιμη μετανάστευση. Ε, τη συζητήσαμε μαζί χθες. Έχουμε δύο, την ε, προστασία των εποχιακών εργαζομένων και τις μεταθέσεις εντός των επιχειρήσεων. Ε, το ένα θέμα αυτό ε, το καλύπτει ο Υπουργό Εργασία τη Δανία, βέβαια, είναι δική του αρμοδιότητα. Ε, αλλά το πρώτο θέμα που αφορά την νόμιμη μετανάστευση και είναι θέμα που θα, θα μας απασχολήσει για πρώτη φορά μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, μας απασχολεί πάρα πολύ και θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος. Ένα άλλο σημείο, το PNR. Το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, θα πω σε λεπτομέρειες. Έχουμε κάποιες ανησυχίες για τις διαπραγματεύσεις εκεί και το ξέρετε. Και το είπατε και εσείς ούτως ή αναφερθήκατε στην παρουσίασή σας. Ε, για το διασυνοριακό έγκλημα και τα δικαιώματα των θυμάτων, ε, εδώ υπάρχει συνένεση, θέλουν εδώ στο Κοινοβούλιο. Αν υπάρξει πρόοδος ε, στα θέματα μας που έχουν κολλήσει, όπως το πακέτο του ασύλου, στο τέλος της Δανέζικης Προεδρίας μπορείτε να τότε μπορείτε να επέρεστε, κοιτάζοντας το παρελθόν, ότι πραγματικά σημειώσατε πρόοδο στην συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Κυρία Βέμπερ, από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας μιλήσουμε στην, εδώ στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ που μας δώσετε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε στα τέλη του 2011 και χθε το απόγευμα. Θα επαναλάβω ουσιαστικά αυτά που είπα και χθε. όλη η ομάδα του, των φιλελεύθερων θα σας ε, στηρίξει. Θέλουμε βεβαίως ε, να πιέσουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας να σημειωθεί πρόοδος σε διάφορα θέματα, αλλά θέλουμε να υπάρχει έτσι, ένα πνεύμα επικοδομητικό στις διαπραγματεύσεις. Θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Ε, από την άλλη βέβαια, σε κάποια θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ, δεν έχουμε άπειρα περιθώρια συμβιβασμού. Θέλουμε να δούμε κάτι αυτό στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Εγώ θέλω να σταματήσω εδώ και να αφήσω άλλους συναδέλφους που είναι ας πούμε εισηγητές σε, επίσημα, σε ευαίσθητα συγγνώμη, θέματα να σας επισημάνουν κάποια σημεία. Καλή τύχη πάντως στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Η κυρία Σαρτζεντίνη από τους Πράσινους. Ευχαριστώ να συνεχίσω κάτι που έλεγαν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Το θέμα της αλληλεγγύης στο πακέτο ασύλου. Ε, το συζητήσαμε χθε, όταν μας συναντήσατε όλου τους συντονιστέ και μου άρεσε αυτή η φράση που είπατε. Την έγραψα μάλιστα. Όλα τα σημαντικά στοιχεία της αλληλεγγύης θα μπουν επιτάπητος. Αύριο και μεθαύριο όταν συναντηθείτε με τους συναδέλφους σας από τα άλλα κράτη-μέλη. Μια τέτοια πρόταση όμως κάποια στιγμή τον Νοέμβριο έφτασε και από τους Πολωνούς. Ήταν προσυπογραμμένη από την Δανέζικη Προεδρία και εκεί αναφερόταν το θέμα της αλληλεγγύης ε, στο πακέτο ασύλου και αφορούσε ουσιαστικά την προστασία των συνόρων, με την αποστολή συνοριοφυλάκων για την προστασία τους. και όχι τους ανθρώπους που χρειάζονται ένα νέο τόπο για να ζήσουν και τις ε, νότιες χώρες που έχουν ε, κατακλειστεί από άτομα τα οποία θα μπορούσαν να ζήσουν κάπου αλλού στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πιθανά θέματα όπου μπορούσε να εκφραστεί η αλληλεγγύη. Πρέπει να τα ξαναδούμε, να τα ξανασκεφτούμε, γιατί πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η λύση και η έκφραση της αλληλεγγύης δεν είναι μόνο η προστασία των συνόρων μας. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σταθώ είναι το θέμα της συνεργασίας. Είπατε ότι θα θέλετε να σπρώξετε την πρόταση για την εντολή για τις ανακρίσεις. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη δικαστική συνεργασία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να ε, δραστούμε. Σας υπενθυμίζω τον, την πράσινη βίβλο που εκδόθηκε στο τέλος του 2011. Ε, βλέπουμε ότι η προδικαστική κράτηση στην Ευρώπη, χρόνος δηλαδή, διαφέρει πάρα πολύ. Και οι εγκαταστάσεις όπου γίνεται αυτή η κράτηση είναι λίγο προβληματικές. Είναι χώρες όπου δεν θα ήθελε κάποιον για, να, για κράτηση εκεί πριν από τη δίκη. Γιατί οι συνθήκες είναι απάνθρωπες, μπορούμε να το θέσουμε έτσι όσο βασίζεται σε αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη η δικαστική μας συνεργασία και όχι σε πρότυπα ε, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στην πρότασή σας, λοιπόν, θα θέλαμε να πιέσετε, να σπρώξετε το θέμα της ε, εντολής για την, τις ανακρίσεις. Ας πούμε, σε ορισμένες χώρες ένα έγκλημα είναι έγκλημα, αλλά σε άλλες όχι. Μπορεί κάποιο να ανακριθεί σε μια χώρα, αλλά όχι σε άλλη. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην αμοιβή εμπιστοσύνη για να χτίσουμε αυτά τα εργαλεία. Ε, όταν, ας πούμε, παραβιάζεται η ιδιωτική σφαίρα, ο ιδιωτικός βίος κάποιου και απειλείται και η ζωή του, ας πούμε. Μπορεί δηλαδή να σε στείλουν σε μια άλλη χώρα ε, για να δικαστείς όπου το σύστημα δεν είναι τόσο αξιόπιστο, όπου η αστυνομία δεν είναι τόσο αξιόπιστη. Ο Ευχαριστώ και καλώς ορίζω τον Δανό Υπουργό και τη Δανέζικη Προεδρία. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα-δύο γενικά θέματα καταρχήν. Καταρχάς, η διεθνής φύση αυτής της ε, Προεδρίας. Τι εννοώ με την λέξη διεθνής. Πρέπει, πρέπει να συζητήσουμε με τη διεθνή κοινότητα αυτή την περίοδο. Ο Δανός υπουργό είχε πάει στη, στη και είχε συζητήσεις και τόνισε τον ενδιαφέρον της Προεδρίας του ε, για τις καλές διατλαντικές σχέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία. Την οικονομική, την πολιτική, Χαίρομαι γι' αυτό και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η τάση και ελπίζω να τελεσφορήσει αυτή η συμφωνία PNR με την της ΕΠΑ. Αναφερθήκατε όπως πρέπει στο γεγονός ότι κάναμε πάρα πολλά εδώ στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Ελπίζω όμως να τελεσφορήσει η δική μου κυβέρνηση και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, αφού περάσαμε από όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία, δέχεται αυτή τη συμφωνία, έχει ένα opt-in. Ως εισηγητής τώρα, τη συμφωνία, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας PNR, εδώ υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες, αλλά παρόλα αυτά ελπίζω να σημειώσουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και ελπίζω να έχουμε καλή σχέση μαζί α, σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, η άποψη της ομάδας μου. Ε, υποστηρίζουμε τις τάσεις και τις προσπάθειες που γίνονται για τη διαφάνεια. Ο Μάικλ Κάσμαν έχουν κάνει πολύ έχει κάνει πολλή δουλειά και άλλοι όμως, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα έγγραφα, είναι διαθέσιμα. Γίνεται μεγάλος λόγος ε, στη διαφάνεια στην πολιτική, για τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή, ας υπάρχει διαφάνεια και στη θεσμική ζωή. Ένας άλλος τομέας είναι ο τομέας του κυβερνοεγκλήματος. Το συζητήσατε. Ο αρμόδιος υπουργός το συζήτησε με, με τους Αμερικανούς στο Τιλαντικό Διάλογο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η μορφή εγκλήματος είναι πολύ σημαντική όσο και οι άλλες ε, μορφές εγκλήματος που αντιμετωπίζουμε. Είναι μια ολένα αυξανόμενη απειλή οικονομικής φύσεως και ελπίζω η Προεδρία θα ετοιμάσει κάποιες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τέλος. Για θέματα ασύλου. Χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη να σημειώσουμε πρόοδο. Υπάρχει ένα δυσανάλογο βάρος σε ορισμένε περιφερειακές χώρες. Και πιστεύω ότι η Προεδρία σας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τη συμφωνία. Το ανέφερα και χθε. Ούτω ώστε να υπάρξει συμφωνία ε, για να αναλάβει ο καθένα την ευθύνη του, ε, με εύλογο τρόπο. Ο καθένα να πάρει το μερίδιο που του αναλογεί. Ε, κάτω από αυτή τη μαγική λέξη τη αλληλεγγύη. Ο κύριος ε, από την ΚΟΕ δεν τον βλέπω που είναι. Ίσως κάποιο άλλο να μιλήσει εξ του. Αν όχι, θα πάμε στους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα εργασίας που ακούσαμε σήμερα το πρωί μου επιβεβαιώνει ότι ε, έχετε το, τα ενία, αλλά δεν αποφασίζετε. Το πρόγραμμα δεν είναι το πρόγραμμα της Δανέζικης Προεδρίας. Είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που, που υπήρχε και θα υπάρχει και μετά τη Δανέζικη Προεδρία. Θα είναι το ίδιο, ακόμα και η Πολωνία να ήταν, το ίδιο θα ήταν, ε, η Κύπρος να ήταν και τα επόμενα χρόνια το ίδιο θα είναι. Ακόμα και αν το Ουσμπεκιστάν είχε την Προεδρία, το ίδιο θα ήταν. Αυτό σημαίνει ότι από τα κράτη-μέλη ε, αφαιρείται η δύναμη, ε, υπάρχουν όλο και περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες, περισσότερη κατάσταση. Ε, και όχι πίσω, δεν πάνε όλοι αυτοί πίσω τι χώρε από τι οποίε ήρθαν, αλλά επε, επανεγκαθίστανται στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσατε για ένα νέο ορισμό των προσφύγων. Φυσικά το χρειαζόμαστε. Αλλά δεν νομίζω θα συμφωνήσουμε επ' αυτού. Νομίζω ότι πρέπει να περιοριστεί σε αυτού που έχουν ε, υποστεί πραγματική δίωξη και όχι σε αυτού που ζουν σε επικίνδυνε χώρε. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Ε, τότε όλο ο πληθυσμό από όλε τι επικίνδυνε χώρε θα πρέπει να έρθει στην Ευρώπη και τότε η Ευρώπη θα βουλιάξει. Αυτοί όμως που έχουν υποστεί διώξεις δεν θα πρέπει να περάσουν από μία ασφαλή χώρα. Γιατί τότε δεν είναι πραγματικοί ε, τούντες άσυλο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αν συνεχίσουν την, το ταξίδι τους, γίνονται οικονομικοί μετανάστες. Μιλήσατε για την απειλή του, της τρομοκρατίας που είναι εισαγόμενοι σε μεγάλο βαθμό. Αναφέρατε κυρίω τον έλεγχο των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών. Αυτή είναι μία από τις πρωτοβουλίε που μου αρέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ατυχέ είναι ότι αναφέρθηκε για πρώτη φορά πριν από αρκετούς μήνες. Μάρτιο ή Απρίλιο του 2011. Θα χρειαστούν μήνες ακόμα πριν περάσουμε στην νομοθεσία για αυτό το θέμα. Βασικά, τους δίνουμε συμβουλές τους ε, τρομοκράτες ε, για το τι θα, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είχαν προγραμματιστεί και ενεργοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα ε, και με εθελοντικές συμφωνίες μαζί με τον κλάδο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν παραβιάσεις αυτής της νομοθεσίας. Όμως, μετά τη Λισαβόνα έχουμε ε, το, τη μόνιμη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έχουμε... Ε, Επίσης, σήμερα το πρωί ακούσαμε ότι γίνονται, ε, έγιναν συναντήσεις ε, στο παρελθόν, αλλά εμείς έχουμε αποκλειστεί. Μετά θα γίνει και μια συνάντηση των συντονιστών. Ε, θα πέσει πολύ γέλιο εκεί. Και εκεί θα υπάρξουν αποκλεισμοί. Πολλοί θα αποκλειστούν από εκεί. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στο Κοινοβούλιο να γίνονται και κλεισμένο των θηρών οι συνεδριάσεις που, που έχουν σημασία σε όλους όσους ανήκουν σε κάποια πολιτική ομάδα. Ακούσαμε έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα. Τώρα θα δώσουμε ξανά το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει και θα τον παρακαλέσουμε να είναι όσο πιο λακωνικός γίνεται, ούτως ώστε να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, γιατί έχω ένα τεράστιο ε, κατάλογο από ομιλητέ. 1,5 λεπτό καθένα θα μιλήσει μετά. Γιατί αλλιώς δεν τα καταφέρνουμε. Ετοιμάστε όλοι σύντομες ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, απαντήστε τώρα όμως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο για τα ενδιαφέροντα ζητήματα που έθεσαν επιτάπητος. Είναι ζητήματα, αυτά που θέσατε, τα οποία είναι στην καρδιά των θεμάτων που μας απασχολούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Και τα θέματα τα οποία θέσατε καταδεικνύουν ότι έχουμε μια κοινή προσέγγιση, θα έλεγα, έναντι αυτών των προβλημάτων, οπότε από κοινού πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται ομαδικά. Θα ομαδοποιήσω τα ερωτήματα για να μην καταχαραστώ το χρόνο σας. Πολύ αναφερθήκατε στο θέμα της αλληλεγγύης. Και τι εννοούμε εμεί ως Προεδρία στο Συμβούλιο με τον όρο αλληλεγγύη. Είναι βεβαίω ένας όρο μια έννοια που ακούγεται συχνά στα ευρωπαϊκά πράγματα. Κατανοώ και συμμερίζομαι το έτοιμά σα θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όταν μιλούμε για αλληλεγγύη. Η Δανική Προεδρία κινείται προ αυτή την κατεύθυνση και αυτό το πρώτο βήμα θα το κάνει αύριο ε, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη και Ιστορικών. Ακριβώ στη μισή διάταξη των Υπουργών είναι το θέμα της αλληλεγγύη. Αναμφίβολα, είναι τεράστια η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια να θέσουμε το πλαίσιο αλλά και το περιεχόμενο της κινητικής πολιτικής εσύλου. Ξέρουμε ότι έχουμε καταληκτική ημερομηνία το 2012 για να συμφωνήσουμε για αυτό το φάκελο. Οπότε η Δανική Προεδρία, αυτό είναι το πρώτο θέμα που θέτει αύριο στην άτυπη Υπουργική Σύνοδο στη ε, στην Κοπενχάγη, θέτοντας το ζήτημα αυτό στην ημερησία διάταξη των Υπουργών. Όταν εμείς ως Προεδρία μιλούμε για αλληλεγγύη, τι έχουμε στο μυαλό μας, πώς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε πρόοδο σε αυτό το τομέα. Πρέπει να εξεύρουμε τρόπους να δημιουργήσουμε ένα πρακτικό πλαίσιο άσκησης ε, της αλληλεγγύης έναν των κρατών μελών που αντιμετωπίσουν ε, τις μεγαλύτερες προκλήσεις, τις μεγαλύτερες πιέσεις. Άρα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια που υπάρχουν ακριβώς για την αλληλεγγύη, άρα μιλούμε για πιο εύκολη χρηματοδότηση και πιο άμεση στήριξη και υποστήριξη των δρατών μελών που αντιμετωπίζουν κατάσταση κρίσης. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα που θα συζητήσουμε αύριο στην Υπουργική Διάσκεψη. Επίσης, η πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης Ασύλου που πλέον έχει πάρει στραγγιωστά, θα πρέπει να συνεπινεγορηθεί βεβαίω από όλα τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι στην πράξη. Πρέπει να δημιουργηθούν πραγματικά οι απαραίτητε εγκαταστάσει για το άσυλο. Να ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρακτικό παράδειγμα τη αλληλεγγύη. Έπειτα πρέπει να υποστηριχθούν οι επιχειρήσει τη Frontex. όπως επίσης να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή δράσης της Frontex. Έπειτα μιλούμε για συνεργασία με τέτοιες χώρες για τους ελέγχου στα σύνορα και εκεί θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και θα πρέπει να συστήσουμε επιτέλους ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα τις ανάγκες που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε έγκαιρα. Έπειτα, πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, Άρα είναι πολύ σημαντικό εδώ να θέσουμε ξανά επιτάπητο στις συμφωνίες επιστροφής. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες να ε, επανεγκατασταθούν είτε στη χώρα προέλευσής τους, είτε κάπου εκεί κοντά, ώστε να μην έχουν ως μόνη διέξοδο τα πολύ επικίνδυνα συχνά ταξίδια προς την Ευρώπη για την εξέβρεση μισοτηρίας. Επίσης, τίθεται πλέον το θέμα της ε, επανακατανομής των ε, μεταναστών, του βάρους των μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών. Είναι ευαίσθητο αυτό το ζήτημα, αλλά αυτά τα έξι σημεία που μόλις ανέφερα θεωρώ ότι αρκούν για να σκιαγραφίσουν ε, την έννοια της αλληλεγγύης έτσι όπως την νοούμε εμείς και πώς την θέτουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Στόχος μας είναι ακριβώς αυτό, να θέσουμε ένα πλαίσιο της πρακτικής έννοιας της αλληλεγγύης, πως πρακτικά δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί ένα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν έντονα αυτές τις πιέσεις και να ενισχύσουμε και τη συνεργασία μας σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα καθώς ανακύπτουν. Όταν μιλούμε λοιπόν για αλληλεγγύη στην πράξη, όπως είπε ο κύριος Μπουστήλ, Αυτή είναι ένας από τους τρόπους που θα προσεγγίσουμε την αλληλεγγύη συγκεκριμένα ξεκινώντας αύριο στην άτυπη υπουργική διάσκεψη στην Κοπενχάγη ώστε να προωθήσουμε έπειτα αυτή τη συζήτηση και να κάνουμε και άλλα βήματα και πιστεύω ότι μπορούμε να εξεύρουμε και τις κατάλληλες λύσεις με αυτόν τον τρόπο. Για το θέμα της διακυβέρνησης Σέγγεν. Πολλά τα σχόλια και πολλές ερωτήσεις που τίθενται. Φυσικά και η Προεδρία μας ανησυχεί για το ζήτημα αυτό. Φυσικά και εμείς θέλουμε την ενεργό και στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις συζητήσεις. Βεβαίως, ε, κατανοείται ότι και εμείς έχουμε μια νέα κυβέρνηση στη χώρα μα και έχουμε ε, μια νέα προσέγγιση για αυτό το ζήτημα της διαχείρισης των συνόρων και της ε, προστασίας της επικράτειας Σέγγεν. Βεβαίως, οι βασικές αρχές που διέπουν την επικράτεια Σέγγεν αποτελούν και τον ακρογωνιαίο λίθο αυτή της προσέγγιση που ακολουθούμε και εμεί. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. θα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την ασφάλεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν ε, σαφείς αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που μας ζητούν να ε, ενισχύσουμε τις προσπάθειες, να κάνουμε κοινέ προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε είναι σαφής η κατεύθυνση. Ο διάλογος με τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που ζητάτε και εσείς, είναι ζητούμενο και για μας. Και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να δώσουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα σε αυτό το τομέα. Θέσατε πολύ και το ζήτημα της Συμφωνίας PNR, της Διαβίβασης Δεδομένων Επιβατών. και πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο ζήτηση είναι η Συμφωνία της Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες εν προκειμένου. Εκ μέρους της Δανικής Προεδρίας θα ήθελα να επισημάνω ότι όταν μιλούμε για την πρόταση PNR ακόμη η πρόταση δεν έχει ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο δεν έχουν κλείσει, οπότε η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι δεν έχει τελική της μορφή. Σε γενικές γραμμές, τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο δείχνουν μια θετική στάση έναντι αυτής της πρότασης για τη διαβίβαση των δεδομένων καταστάσεων επιβατών. γιατί είναι κάτι αναγκαίο για τη λειτουργία των αρχών επιβολής της τάξης και του νόμου. Οι διεκτικές αρχές θεωρούν ότι είναι ένα ουσιώδες, απαραίτητο εργαλείο για ανταλλαγή των δεδομένων PNR για να μπορούν να διερευνήσουν πιο αποτελεσματικά μία σειρά εγκληματικών δραστηριοτήτων. Είναι ένα θέμα που συζητήσαμε ήδη από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την ε, Προεδρία ε, στην πρώτη επίσημη ε, σύνοδο που έγινε στην Κοπενχάγη για την ανάληψη Προεδρίας, αλλά και σε επαφές στις άτυπες που είχα μαζί σας πριν τα Χριστούγεννα. Για μας, στο Συμβούλιο, το PNR είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να εξεύρουμε αποτελεσματικέ λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως και θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας εν προκειμένου και βεβαίως πρέπει να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία. Όμως, αυτό που είπα ευθύς εξ αρχής ήταν ότι, και εγώ το είπα δηλαδή, ότι η η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής δεν σημαίνει εν λευκό επιταγή και καταπάτηση ατομικών ε, και πολιτικών ελευθεριών. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο. Έπειτα, ε, ένα άλλο θέμα είναι η πρόταση για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Θέσατε και κάποιες ερωτήσεις για αυτό το ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι η διαφάνεια που θα πρέπει να διέπει τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης είναι ε, ουσιώδες στοιχείο που χαρακτηρίζει και τη δική μας παράδοση αυτή τη στιγμή ε, το Δανικό Κοινοβούλιο συζητά ένα τέτοιο πακέτο ε, νέων νομοθετικών ε, προτάσεων. Προσβλέπουμε λοιπόν στις, στη συζήτηση της, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο με στόχο να βρούμε την πλέον ρεαλιστική λύση για να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία και για αυτό το φάκελο. Είναι προφανές πάντως ότι όταν μιλούμε για εθνικές διοικήσεις δεν μιλούμε ακριβώς για το ίδιο πράγμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν εθνικές ιδιαιτερότητες. Και άρα και οι προσεγγίσεις μας διαφέρουν σημαντικά. Κατά την εξέταση λοιπόν αυτής της πρότασης πρέπει να δεχτούμε τις εθνικές παραδόσεις ε, ε, και ε, αντιμετώπιση του θέματος της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και την έννοια της διαφάνειας. Και αν με επιτρέπει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση θέτοντας ε, το ζήτημα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η ηλεκτρονική επιλογή οι εγκληματικές ενέργειες μέσα στο διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη και σήμερα και θα παραμείνει και στο μέλλον. Η Δανική Προεδρία έχει προβλέψει ένα σεμινάριο στην Κοπενχάγη για το ηλεκτρονικό έγκλημα και θα λάβει χώρα συγκεκριμένα το Φλεβάρι. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην φάση των ερευνών θα έρθουν και θα μιλήσουν σε αυτό το σεμινάριο άνθρωποι που ασχολούνται πρακτικά με αυτή τη φάση της έρευνας, της διερεύνησης τέτοιων εγκληματικών ε, πράξεων μέσα στο διαδίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός φάκελος αυτός, γι' αυτό ε, είναι τόσο ψηλά στις προτεραιότητες μας. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο οδηγίας για την επίθεση στα συστήματα πληροφορική, στα συστήματα IT, θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόταση και ελπίζουμε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ελπίζουμε να έχουμε και ένα εργαστό διάλογο και για αυτό το θέμα. Και τέλος, αν μου επιτρέπει και πάλι ο Πρόεδρος, για την κυρία Σαρτζεντίνη αν μου επιτρέπετε και ελπίζω να πρόφερα και ορθά το όνομά σας. Το θέμα που θέσατε είναι θεμελιώδες. Η αμοιβή εμπιστοσύνη, κατά με, είναι θεμελιώδε ζήτημα. Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όταν μιλούμε για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών μελών είναι θεμελιώδε στοιχείο. Γι' αυτό και μέσα στα πλαίσια τη αμοιβαίας εμπιστοσύνη εντάσσεται και η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνα. το περίφημο ΕΙΟ. E Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το κατάλληλο πεδίο για να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα συστήματα επιβολή τη τάξη και του νόμου μεταξύ των κρατών μελών. Και η αμοιβή είναι θεμελιώδη στοιχείο για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις τεράστιε προκλήσεις που έχουμε. Παράδειγμα, να σας δώσω. Υπάρχει ένα σύγχρονο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πρέπει να κλείσουν οι προτάσεις για τα δικαιώματα των κατηγορουμένων για εγκληματικές πράξεις και την πρόσβασή του συγκεκριμένα σε ε, συνήγορο. Πιστεύω ότι υπάρχει ήδη κατάλληλη βάση για να συνεχιστούν οι καλές συζητήσεις και για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Πρόεδρος, ο Υπουργός άκυξε ήδη τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα που θα αποτελέσουν ε, και τα θέματα που ασχολήσουν την Προεδρία και αφορούν και την Επιτροπή μα. Αναφέρθηκε και στο σεμινάριο για το ηλεκτρονικό έγκλημα που θα λάβει η χώρα στην Κοπενχάγη το Φλεβάρι. Τώρα θα ξεκινήσω ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να εμείνετε σε θέματα που δεν ετέθησαν ήδη στον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Σας παρακαλώ πολύ να καταβάλετε κάθε προσπάθεια να μην ξεπεράσετε το 1,5 λεπτό. Έχω κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών Κοέλιο, δύο Ford, Mrs. Romero Lopez, Mrs. Alfano, Mr. Κλείνει ο κατάλογος. 15 αγορητές, 1,5 λεπτό έκαστος και θέλω να υπενθυμίσω και στον Υπουργό ότι είναι πολύ σημαντικό και εκείνος να είναι συνοπτικός στην ε, δεύτερη του απάντηση. Ο κύριος Κοέγιο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του και για την τοποθέτησή του. Εκτίμησα ιδιαίτερα τα λόγια που είπατε για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τον αναφορά σα στον κεντρικό ρόλο που έχει ο χώρο Σέγγεν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ελευθερία κυκλοφορία και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια ασφάλεια. Υπ' αυτή την έννοια, χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα αξιολόγηση Σέγγεν. Όπω γνωρίζετε πολύ καλά, διάφορα κράτη-μέλη προτιμούν να μειώσουν το πήγη της φιλοδοξίας της προτάσεις τους και επιλέγουν μία άλλη λύση που θα είναι αυτή που δεν θα επιτρέψει τη συναπόφαση στο Κοινοβούλιο. Οπότε ρωτώ συγκεκριμένο σε εσά. Ω Υπουργό τη Δανία και ω ε, εκπρόσωπο Προεδρία, συμφωνείτε με αυτόν τον προσανατολισμό, ή θα προσπαθήσετε να διαφυλάξετε την απόφαση για το Κοινοβούλιο. Δεύτερη και τελευταία ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για το SIS, κατά τη γνώμη της Προεδρίας, θα μπορεί να διατηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα ή υπάρχουν προβλήματα που σας υποχρεώνουν να πανεξετάσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα και άρα θα καθυστερήσει για μια ακόμη φορά η θέση ισχύ αυτού τόσο σημαντικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χέντ, δεν είναι εδώ. Η κυρία Ρωμένο Λόβεθ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Μπόσκοτ εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα που αφορούν το πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Βλέπω ότι έχετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και σας εύχομαι καλή επιτυχία, διότι το ζήτημα του ασύλου και ένα κοινό σύστημα ασύλου είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα που α, ήδη ξέρουμε από την εμπειρία και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ότι παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Ήδη πολλέ οδηγίε δεν υιοθετηθήκαν έω σήμερα και ούτε γνωρίζουμε ακριβώ τι θα ήταν ένα κοινό σύστημα ασύλου. Και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου στην Μάλτα μόλι τώρα ξεκίνησε να λειτουργεί. Μέχρι πού πιστεύετε ότι μπορεί να πάει και τι μπορεί να καταφέρει η Δανική Προεδρία, διότι δεν είναι μόνο ο μηχανισμός έγκρισης προειδοποίησης της Πολωνικής Προεδρίας, αλλά και τα κέντρα κράτηση των μεταναστών είναι κάτι που πρέπει να σας απασχολήσουν. Όπως και τα κράτηση των ετούτων άσυλο. Είναι σαφές ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζεται σήμερα στη Βόρεια Νιγηρία και με την δίωξη των χριστιανών όπως και στη Σομαλία μας αναγκάζει να επαναθεωρήσουμε τον ορισμό της έννοιας μη ασφαλούς χώρας. Πρέπει να ορίσουμε πλέον διαφορετικά την έννοια της μη ασφαλούς χώρας και να ξεφύγουμε από τη σύμβαση της Γενέβης. Διότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, που εγκαταλείπουν τη χώρα τους και δεν εμπίπτουν στον ορισμό της σύμβασης της Γενέβης. Δεύτερο ζήτημα τώρα που θέλω να θέσω και αφορά το πακέτο για τα θύματα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε στατιστικά στοιχεία για τα θύματα βίας α, και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε γυναίκες και παιδιά. Διότι, ναι, μεν γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά έρχονται καθυστερημένα. Θα μπορούσε η Eurostat να στηλέξει δεδομένα ώστε να κατανοήσουμε πόσο ευρύ είναι αυτό το φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή και να καταλήξουμε σε μια σχετική στρατηγική. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λάτφορντ και παρακαλώ, 1,5 λεπτό είπα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ είναι η συζήτηση για το PNR και τις ανταλλαγέ ε, ανταλλαγές πληροφοριών προσωπικών δεδομένων. Αυτό λοιπόν το θέμα. Δεν αφορά μόνο, πιστεύω, επιβάτες ε, πτήσεων, λίστες δηλαδή επιβατών πτήσεων. Όταν κάποιος ε, προσδιορίζεται ότι πρέπει να υποστεί δεύτερη ε, εξέταση, δεύτερη, δεύτερο πέρασμα από τα μηχανήματα, επειδή υποτίθεται ότι έχει χαρακτηριστικά ε, λαθρεμπόρων, ναρκωτικών κτλ. Ε, αυτομάτως μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και σε κάποιους, οι οποίοι μπορεί να χαρακτηρίζονται ως υπόπτη τρομοκρατίας, όπως έγινε με κάποιον ο οποίος ε, ονομαζόμενος Μπενιέ Μοχάμετ ήταν στην ίδια πτήση μαζί με έναν πατήλα ο οποίος καταδικάστηκε για τρομοκρατική δραστηριότητα χωρίς όμως να έχει βάλει βόμβα μέσα στο αεροπλάνο για άλλου τύπου τρομοκρατική δραστηριότητα όμως ο πρώτος ο οποίος απλώς συνευρέθη τυχαία ε, ως επιβάτη στο ίδιο αεροπλάνο με τον ε, κατηγορούμενο Παραπέφθηκε παραπέμφθηκε στις φυλακές του Γουαντάναμο όπου, όπου ε, υπέστη φοβερά βασανιστήρια. Το ίδιο έχει συμβεί και σε άλλους που τυχαία βρίσκονται έτσι ε, γιατί τους χαρακτήρισαν ως υπόπτους κάποιοι και κατά τρόπο τελείως αδικαιολόγητο. Εάν λοιπόν αυτές οι πληροφορίες αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής χωρίς καμία βάση ουσιαστική και κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι να ε, ε, να χαρακτηριστούν διαπαντός ως ύποπτοι για ο,δήποτε έγκλημα, τότε τους έχουμε, ε, έχουμε τεράστιο πρόβλημα ως προς την των δικαιωμάτων τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κυρία Φλότρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Λάτφορντ ε, μίλησε για συγκεκριμένες υποθέσεις ε, στον τομέα της ε, πάταξης τρομοκρατίας και τις, τα μέτρα που λαμβάνονται. Εγώ θα ήθελα, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξαναρχίζει τις προσπάθειές του μετά τις εργασίες του 2006-2007, προκειμένου να ρίξουμε φως στο ζήτημα της έκτακτης ή παράνομης παράδοσης ε, από τις Ηνωμένες, στις Ηνωμένε των Ηνωμένων με τις πολύ σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων που διαπιστώθηκαν τότε από το Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε λοιπόν εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζουμε κατά πόσον το Συμβούλιο, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, Κατά πόσον λοιπόν σκοπεύετε, δεδομένου ότι και η ε, Προεδρία σας ε, συμπίπτει χρονικά 100% με τις εργασίες του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να εκδώσει τις θέσεις του, να δημοσιεύσει τις θέσεις του προς το τέλος της δικής σας θετίας. Εάν λοιπόν σκοπεύετε, όπως έλεγα, προκειμένου να κάνετε, να κάνετε αυτό που οφείλετε, δηλαδή να ρίξετε άπλετο φως στην υπόθεση αυτή για όλους, να προχωρήσετε. Σε ποιο βαθμό, ερωτώ, είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε μαζί μας, κύριε Υπουργέ. Το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εννοείται κύριε Υπουργέ ότι σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και να πάω κατευθείαν στα ερωτήματά μου. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Ρομέρο Δηλαδή, τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, θα υπάρξει συμφωνία τελικά. Να σα υπενθυμίσω ότι στο πρόγραμμα Χάκε και την ε, σχέδιο δράση υπήρχε μία δέσμευση για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 2010. Ακόμη περιμένουμε. Λοιπόν, εγώ εκφράζω την εμπιστοσύνη μου προ τη Δερική Προεδρία. Δεύτερον, δεν άκουσα τίποτα στην προσέγγιση σα σχετικά με τον νέο ε, κανονισμό για την Europol. Πρόγραμμα Στοκχόλμη ε, και σχέδιο δράση. Και ένα περίπλοκο ερώτημα. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε. Θα κατανοήσω αν δεν μου απαντήσετε. Αλλά θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει το ζήτημα που θα θέσω. Αναφέρω στο κανονισμό 539 του 2001 και ένα κάπως δηλητηριώδες ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Μια τρίτη χώρα επιβάλλει υποχρεώσεις θεωρήσεων είναι κράτος μέλος. Σας παρακαλώ τουλάχιστον να μου δώσετε το να με παρακολουθείτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, όταν, όταν μια τρίτη χώρα επιβάλλει υποχρεώσεις θεωρήσεων σε ένα κρατός μέλος, εσείς, η, η ιδανική προεδρία, συμφωνείτε με μια αυτόματη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια κοινή αυτόματη απάντηση. Είναι νομικά εφικτή μια τέτοια κοινή αυτόματη απάντηση. Ξέρω ότι η απάντησή σα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη και περίπλοκη σε πολιτικό επίπεδο. Οπότε θα κατανοήσω αν δεν μου απαντήσετε αυτή τη στιγμή. Όμως παραλαμβάνω πολύ σημαντικό ζήτημα και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα σε λιγάκι. Θα ήθελα να εμβαθύνετε επί του θέματο, ώστε να έχουμε κι εμεί μια εικόνα για το ποια είναι η στάση τη δανική Προεδρία. Χτες, οι συνεργάτε σας, στην επαφή που είχαμε, μας ε, έδωσαν ένα δείγμα πολύ επαγγελματική γραφής και ότι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Το αναφερθήκαμε στον κανονισμό του Συμβουλίου 539 κάθετος 2001 και αφορά τον κατάλογο εκείνων των χωρών οι υπήκοοι των οποίων θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή του θεώρηση κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιοι εξαιρούνται από αυτή την απέτηση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Σκεφτείτε το για να απαντήσετε στον κύριο Δία Ντεμέρα. Προχωρούμε τώρα στον κύριο Ένσιο. Ενάμιση λεπτό. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să felicit și eu pe domnul ministru și de asemenea președinte. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό και τη Δανέζικη Προεδρία για τους στόχους που έχει θέσει, που είναι πολύ φιλόδοξοι. Και γιατί δείχνει ανοιχτό πνεύμα για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή μας των Δημοσίων Ελευθεριών. Θα σας υποστηρίξουμε, εάν θέλετε τη βοήθειά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε μαζί τα πιο σημαντικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία μόνη έκκληση θέλω να σας απευθύνω. Ελπίζω κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να τα καταφέρετε, να πείσετε ένα κράτος μέλος που αντιτίθεται σε ένα φάκελο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ούτως ώστε να ενταχθούμε στο χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ τον ε, Υπουργό. Θέλω να σταθώ στο τελευταίο τμήμα Υπάρχει μια πολύ ανησυχητική κατάσταση στην Ουγγαρία. Εσείς θέλετε να ανοίξει η διαδικασία του άρθρου 7, όπως πρότεινε ο Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργο, για το οργανωμένο έγκλημα. Ήμουν εισηγήτρια για, για το θέμα αυτό και το Δεκέμβριο έστειλα ε, έγγραφο, αντίγραφο στο γραφείο σας. Τι δέσμευση θα πάρετε για την, το οργανωμένο έγκλημα και τη μαφία στην Ευρώπη. Στις 12 και 13 Μαρτίου βλέπω ότι θα υπάρξει ένα σεμινάριο της Προεδρίας σας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτό το θέμα, για αυτό το σεμινάριο. Σας τα ρωτάω αυτά γιατί σήμερα το απόγευμα στο... στις Βρυξέλλες θα παρουσιάσω αυτό το βιβλίο το οποίο εξηγεί και αναφέρει ε, ένα τμήμα από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής που λέει ότι το, το έγκλημα αυτό ε, κοστίζει ε, εκατοντάδες εκατομμύρια ε, ευρώ για τη διερεύνησή του σε διάφορες χώρες, Ισπανία, Βέλγιο κτλ. Συγγνώμη, από μυστικές υπηρεσίες εδώ στο Βέλγιο. Domnule președinte, <clears throat> domnule ministru, subiectul intervenției mele... Έχει αναφερθεί αυτό που ήθελα να πω εγώ. Μιλάω για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Υπάρχει υποστήριξη της Πολωνικής και Ουγγρικής Προεδρίας για, αυτό το, για αυτή την ένταξη, αλλά δεν είχαμε αποτελέσματα. Ελπίζουμε να υποστήριξετε κι εσείς την ένταξή μας στο χώρο Σέγγεν. Θα δείξετε την ίδια... Αν όμως κάνετε τα ίδια με τις προηγούμενες προεδρίες θα γίνει τίποτα. Νομίζω ότι η Ολλανδία που αντιτίθεται θα πρέπει να καταλάβει ότι ε, τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη και η ίδια η Ολλανδία πρέπει να σεβαστεί τις συνθήκες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να δεχτεί το γεγονός ότι αυτές οι δύο χώρες πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεκτημένο Σέγγεν. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να πάρει μια απόφαση για την ένταξη των δύο χωρών. Ε, ποια είναι η άποψή σα, κυρία Αντζελίλη, μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ εσά και την Δανέζικη Προεδρία για το φιλόδοξο πρόγραμμα. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που ακούσαμε από συναδέλφου. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα μόνο. Εσείς υπογραμμίσατε τη σημασία της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού χώρου ελευθεριών, πραγματικών ελευθεριών για τους πολίτες. Μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών είναι και τα παιδιά. Και όπως τα ξέρετε βεβαίως, με την αύξηση της ε, κυκλοφορίας των προσώπων υπήρξε αύξηση αναπόφευκτη, αλλά και θετική, έτσι, των γάμων, Μερικές φορές όμως υπάρχουν, προκύπτουν και χωρισμοί και διαζύγια. Μερικές φορές όταν, γίνεται, όταν υπάρχει ένα διαζύγιο α, δημιουργούνται προβλήματα, διδικίες κτλ. Και δυστυχώς την πληρώνουν τα παιδιά. Γιατί ενδεχομένως ένας γονέας απάγει το παιδί και το στερεί από τον άλλο γονέα. Και δεν ε, επιτρέπει στο παιδί να ασκήσει το δικαίωμά του για σχέσεις και με τους δύο γονείς, όπως προβλέπετε και από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και πάω στο ερώτημά μου. Η Δανία δεν έχει ακόμα υιοθετήσει τον κανονισμό 2α για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε ό,τι αφορά την γονική ευθύνη. Επομένως, δεν συμμετείχε δεν συμμετέχει στη δικαστική συνεργασία στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την, τα θέματα των ανηλίκων. Σας παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε αυτό το ερώτημα. Ο κύριος Μπορσελίνο. Η κυρία Μπορσελίνο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτή τη συζήτηση. Είμαι εισηγήτρια για την ε, στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη. Είπατε σημαντικά πράγματα και για την ασφάλεια ε, που πάει χέρι-χέρι με την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν αφορά μόνο τις ε, χώρες μέλη, αλλά η αλληλεγγύη αφορά, είναι η στάση και προς τα άτομα. Μιλάτε για το, το πακέτο για τα θύματα, για την μετανάστευση, για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ λεπτά και ευαίσθητα. Εδώ σε λίγο θα μιλήσουμε ε, για την αποστολή που κάναμε στη Λαμπεντούζα στη Σικελία για να δούμε τα θέματα της μετανάστευσης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, λόγω αυτών των εμφάσεων που σας ανέφερα, να θυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων που θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα μια και είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά αξίζει να το ξαναπούμε και να βάλουμε έμφαση εκεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Υπουργό για τη σημερινή του παρουσία στην Επιτροπή μας. Ως εισηγητρία στην Επιτροπή μας για την οδηγία, για την στήριξη, προστασία και δικαιώματα των θυμάτων, διαπιστώνουμε ότι αυτή η οδηγία είχε, είχε τύχει πολύ καλή υποδοχή εξ αρχής και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν θέσει πολλές ελπίδε στην οδηγία αυτή και δεν πρέπει να σου απογοητεύσουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας τάση του θέματο, αλλά θέλω να διευκρινίσετε το εξή. Όταν είπατε ότι αυτή η οδηγία θα υποστηριχθεί υπό την αίρεση της παρούσας οικονομικής κατάστασης. Τι ακριβώς εννοείται. Όταν μιλάτε για την παρούσα οικονομική κατάσταση, τι εννοείται. Ότι θα μειωθεί το επίπεδο υποστήριξης των θυμάτων χρηματικής δηλαδή στήριξης. Επίσης θέλω να επαναλάβω ότι η Δανική Προεδρία έχει ήδη δεσμευτεί να υποστηρίξει τα δικαιώματα των θυμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σε ευχηθώ πάντως κάθε επιτυχία της Προεδρίας σας για τα καλύτερα αποτελέσματα και ελπίζω να μην μειώσω τον πύχη σε σχέση με τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την οδηγία για τα θύματα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τηρώντας το κώδικα θετολογίας Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Ευχαριστώ τον Υπουργό, ε, μάλλον εκ των προτέρων, για την προσπάθειά του να είναι τόσο συνοπτικό στην απάντησή του, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα σημεία. Έχετε το λόγο. Øh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις οι οποίες είναι θαυμάσιες, πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ακολουθήσω την συμβουλή του Προέδρου, λοιπόν, και θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ λακωνικός. Ούτως ή άλλως θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα. Γιατί, όπως σας είπα, θέλω πραγματικά να υπάρχει ανοιχτό και τακτικός διάλογος μεταξύ μας. Μου θέσανε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο χώρο του Σέγγεν. Θέλω να τονίσω το εξής. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, τα συγκεκριμένα, εγώ τουλάχιστον και η Προεδρία, επιθυμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί στη διαδικασία που αφορά αυτή την πρόταση για το Σέγγεν. Αυτό είναι προφανές. Η κυρία Λόπες έθεσε ένα ερώτημα για το πακέτο που αφορά το άσυλο και για το πακέτο για τα θύματα. Για το πακέτο για τα θύματα θα σας μιλήσω σε λίγο. Για το σύστημα ασύλου καταρχήν και τις υποχρεώσεις που έχουμε. Στα πλαίσια αυτού του πακέτου. Θα κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός αν ε, εγκύψουμε στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου πραγματικής και πρακτικής αλληλεγγύης, για να το πω έτσι. Σας μίλησα ήδη για τα έξι σημεία όταν έκανα την αρχική μου παρουσίαση. Δηλαδή, την προσπάθεια δημιουργίας μιας πραγματικής και πρακτικής αλληλεγγύης που θα περιλαμβάνει αυτά τα έξι σημεία, που κατά την άποψη τη Δανική Προεδρίας θα μας επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Η συζήτηση μάλιστα θα ξεκινήσει αύριο το πρωί στην Κοπενχάγη στα πλαίσια αυτής της άτυπης συνάντησης. Εμείς η Δανέζικη Προεδρία ε, θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουν οι συζητήσεις και να βρούμε ένα πλαίσιο για μια πραγματική, για μια απτή και πρακτική αλληλεγγύη. Ένα άλλο ερώτημα ήταν αυτό που έθεσε η κυρία Λάτφορντ. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας, κυρία μου. Ε, οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν τις πληροφορίες που δίδονται στα πλαίσια του PNR, του Passenger Name Record. Έγινε μια διαπραγμάτευση μεταξύ ημών και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πιο γενικά αφορά το θέμα αυτό την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών, των ευαίσθητων στοιχείων. Όταν μιλάμε για, κρά... για τήρηση κάποιων στοιχείων που αφορούν προσωπικές πληροφορίες, θα πρέπει να ξέρουμε ποιε είναι οι πληροφορίε που κρατάμε και πώς τις κρατάμε αυτές τις πληροφορίες, ε, με έναν τρόπο αναλογικό. Αυτή η αναλογικότητα είναι το βασικό θέμα της συζήτηση. Και ελπίζω να βρούμε λύση με τις Ηνωμένε Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα δεδομένα PNR. Είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων, λεπτών, προσωπικών, ευαίσθητων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την προστασία τους. Προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Η κυρία Φλότχα μίλησε για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι και δική, μας ευχή και δικός μας διακαής πόθος αυτή η συνεργασία. Δεν θα πρέπει να έχετε καμία αφιβολία γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το νέο κανονισμό για τη Europol. Ακούστηκε μια ερώτηση επίσης. θα πρέπει να δούμε τη θέση της Κομισιόν. Και εν συνεχεία εμείς θα πάρουμε θέση σε σχέση με την θέση της Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα για να σας πω ποια θα είναι η θέση μας. Δεν μπορώ να δεσμευτώ από τώρα. Ούτω ή άλλω είμαστε, αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι είμαστε έτοιμοι για διάλογο. Ανοιχτό και επικοδομητικό. Δεν μπορώ επίσης να προδικάσω το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θα πετύχουμε, αλλά θα παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως φαντάζεστε. Εν συνεχεία. Πολλοί από εσά. Μίλησαν για την ε, ένταξη της Ρουμανίας και Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν. Είναι πολύ σημαντικό ειδικά τώρα, όταν προτιθέμεθα να λάβουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Προεδρία μας πιστεύει ότι δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο, νομικό κόλλημα που εμποδίζει τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία να ενταχθούν 100% στο χώρο Σέγγεν. Θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά το ότι, ότι, το ότι η συνεργασία μας θα πρέπει να βασίζεται σε διαφανείς και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Για να είναι πραγματική αυτή η συνεργασία. Δεν πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια συνεργασία ε, η οποία θα οδηγήσει σε ένα σύστημα πολλαπλών ταχυτήτων σε δύο μέτρα και δύο σταθμά ή τρία μέτρα και τρία σταθμά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Η κυρία Αλφάνα, Αλφάνο μάλλον, μίλησε για την Ουγγαρία και το Αρθεφτά. Και όπως είπατε, κύριε Αλφάνο, αυτό το θέμα έχει ξανασυζητηθεί με διάφορους υπουργούς. Και η Κομισιόν στάθηκε σε τρεις παραβιάσεις της Ουγγαρίας έναντι των συνθήκων μετά την ε, τροποποίηση του συντάγματος της. Είναι ένα κρίσιμο θέμα αυτό, φυσικά. Και εμείς ως Προεδρία θα είμαστε σε συνεχή διάλογο με την Κομισιόν για το σημείο αυτό της Ουγγα... Ουγγαρίας. Εν συνεχεία μιλήσατε για την, για την οργανωμένη εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα. Μιλήσατε για ένα βιβλίο Τώρα, από την εμπειρία τη δική μου, από αυτά που ξέρω, από τη Δανία. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσο πιο στενή είναι η συνεργασία μεταξύ των αρχών, δηλαδή της, των φορολογικών αρχών, των διοκτικών αρχών, μπορούμε έτσι να αυξήσουμε την, την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Και εδώ στην Ευρώπη το, το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Ε, στενή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αρχών. Αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να προβλέψουμε, να προλάβουμε τα αποτελέσματα του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, είναι τεράστια πρόκληση. Πάντω η στενή συνεργασία δίνει αποτελέσματα. Ε, καταπολεμούμε συμμορίε, οργανώσει κτλ. Ε, συνεργασία των αρχών στο εσωτερικό τη χώρα αλλά και διασυνοριακά. Ειδικά των αρχών που διεξάγουν την έρευνα. Αυτές οι αρχές πρέπει να συνεργάζονται γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Κύριε Αντζελίλη έθεσε ένα ερώτημα για τα παιδιά. Εμείς στην Δανία δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά προβλήματα. Ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα. υπήρξε ένα τελευταίο ερώτημα για το πακέτο για τα θέματα και τα δικαιώματά τους. Ελπίζω να συνεργαστούμε καλά. για το πακέτο αυτό. Η Πραδία θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για την Ευρώπη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, παράδειγμα από τη Δανία. Έχουμε opt-out σε νομικό επίπεδο. Για, αν η Δανία, ας πούμε, διώκεται, την τυρανά ένας βίος σύζυγος, ας πούμε, στη Γερμανία, μπορεί στη Γερμανία να πετύχει μια απόφαση κατά του συζύγου της. Αλλά όταν επιστρέψει στη Δανία θα χάσει αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από το, να ξεφορτωθούμε αυτό το opt της Το θέμα των, των δικαιωμάτων των θυμάτων και το θέμα της οικονομικής πραγματικότητας που περιβάλλει αυτά τα δικαιώματα δεν αφορά μόνο τα ίδια τα θύματα. Συνδέεται και με άλλες προτάσεις το πακέτο αυτό για τα θύματα. Μην ξεχνάμε την οικονομική κρίση στην Ευρώπη πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα μέσα και να τα αντιπαραβάλουμε με τις ανάγκες που έχουμε στην Ευρώπη. Ως πρόεδρος θα κάνω τι μπορώ, ούτως ώστε να περάσουν αυτές οι προτάσεις. Ελπίζω ότι μαζί θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Ελπίζω να φτάσουμε πιο κοντά στη λύση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ επωφελέ για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ σε ευχαριστώ και σα εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία Σα Ευχαριστούμε για την ακρίβεια, για τη λεπτομέρεια με την οποία προσπαθήσατε να απαντήσετε σε κάθε ερώτημα που ακούστηκε και προσβλέπουμε σε μια περαιτέρω ενίσχυση τη συνεργασία μα αυτό το εξάμεινο. Βεβαίω, θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε για να εκφράσουμε τη συνεργασία μα με τη Δανική Προεδρία ειδικά το εξάμεινο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και κάτι που. Α, η κυρία Ρομέρο θέλει να θέσει κάτι. Παρακλείστε πάρα πολύ σύντομη όμω. Κύριε Ρομέρο, δεν ξέρω αν μήπως ξεχάσετε να μου απαντήσετε στο δικό μου ερώτημα. Δεν είναι ερώτηση που αφορά αύξηση του προπολογισμού. Μίλησα για στατιστικά δεδομένα για τα θύματα βίας. Μπορείτε να κάνετε κάτι για να συλλέξουμε τέτοια στατιστικά δεδομένα στη Eurostat. Το θέσαμε το ερώτημα στου προηγούμενους υπουργού δικαιοσύνη ε, που είχαν την Προεδρία. Πόσα θύματα βίας έχετε στη χώρα σας. Είναι πολύ σημαντικό να ε, στατιστικά στοιχεία. Ναι, ναι, να απαντήσει ο υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία διαθέσιμα. Το πακέτο για τα θύματα ε, δείχνει πώς μπορούμε, μας δείχνει το δρόμο αν θέλετε, για να δούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα πρακτικά. Όμως, σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε και για ειδικού είδους βοήθεια σε όλα τα επίπεδα για τα θύματα, ε, για να μπορούμε να τους ε, δίνουμε πρακτική προστασία. Ευχαριστώ, λέει Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να αποδείξουμε ότι θέλουμε να εργαστούμε από κοινού για να προωθήσουμε όλους τους φακέλους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να ζευτεί με επιτυχία Προεδρία της Δανίας, στην οποία βεβαίω ευχόμεθα κάθε επιτυχία. Σε ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. So, we keep working. Now we move to the following point, which is an information. Να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι ενημερωτικό για τη Σικελία, αποστολή στη Λαμπετούσα, που έκαναν κάποια μέλη της Επιτροπής Κολέγκα με επικεφαλή στην κυρία Βίκστρομ, επικεφαλή της ε, ε, αντιπροσωπείας μας ε, στην επίσκεψη στην Λαμπετούσα για να γίνει μια επιτόπια εξέταση της μαζικής εισρωής μεταναστών. Έλαβε χώρα αυτή η επίσκεψη 24 και 25 Νοεμβρίου Παρακαλώ κύριε Βίξτρομ να είσαστε σύντομοι για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το ε, κενό που πρέπει να καλύψουμε γρήγορα. πείτε, Πρόεδρε, να περιμένω αν θέλετε μερικά δευτερόλεπτα για να σταματήσει η φασαρία στην αίθουσα. Πρόεδρος, ναι, να θυμίσω σε όλους όσους εγκαταλείπουν την αίθουσα, ήσυχα παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βίξτρομ, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους ε, για την προσπάθεια να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα για σήμερα. Ε, υπάρχει ήδη μια σύντομη σύνοψη των εντυπώσεών μας μετά την πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στη Σικελία και στη Λαμπετούσα 24-26 Νοεμβρίου 2011. Θέλω και πάλι να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου στην Μαρίαν Χέλενα από τη Γραμματεία, του Συμβούλου πολιτικής που μας συνόδευσαν και τους εννέα συναδέλφους στην εκπροσωπεία. Τα πρακτικά αυτής της επίσκεψης τα έχετε ήδη λάβει και απεστάλησαν και στο γραφείο μετάφρασης. Θέλω να σχολιάσω τώρα το τι αποφασίσαμε να κάνουμε ως follow-up Είχα μια επαφή με εκπροσώπους της ε, μόνιμης Ιταλικής Επιδοσοπίας, απέστειλε και μια επιστολή στις Ιταλικές Αρχές και δίνημα την σχετική αυτή επιστολή σε όλους σας. Γνωρίζω, σε ό,τι αφορά τη μόνιμη προσωπία της Ιταλίας, είναι έτοιμοι να μας δώσουν μια ε, επίσημη απάντηση, την οποία θα λάβουμε σύντομα. Μόλις λάβουμε την επίσημη απάντηση της αντιπροσωπείας, θα σας την διανύμουμε σε όλη την Επιτροπή εντάχει να πω, γιατί δεν θέλω τώρα να διατρέξω το κείμενο, τα πρακτικά είναι αρκετά ενδελεχή, αλλά με το που γυρίσαμε στις Βρυξέλλες σας ε, δώσαμε μια πρώτη εντύπωση, σας δείξαμε φωτογραφίες κτλ. Αν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να σχολιάσετε, παρακαλώ να με ρωτήσετε. Σας προτείνω να διαβάσετε πρακτικά, τα οποία θα μεταφραστούν και σύντομα και θα λάβετε τη μετάφραση. Μετά τη μετάφρασή τους θα υιοθετήσουμε τα πρακτικά στην συνεδρία της Επιτροπής μας το Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτά, Πρόεδρε, και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίξτον. Για την έκθεση και τώρα ας ακούσουμε τους συναδέλφους. Για Κολίνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, η επίσκεψη στη Σικελία, στο Τράπεντο, ε, κράγατα, τη Λαμπετούσα και στο Παλέρμο, και το μήνυμα, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία να έρθουμε σε κοντινή επαφή με τους ντόπιου, όπως ε, επίσης και η στενή επαφή με τους μετανάστες εκεί. Διάβασα τα πρακτικά της συναδέλφου της κυρίας Γουίξτρομ Θα προτιμούσα πάντως ότι πέρα από μια απλή ενελεχή ε, περιγραφή ε, των τετεκτονωμένων με απέραντη σχολαστικότητα όλων όσων δημήθησαν σε αυτή την επίσκεψη, θα ήλπιζα να υπήρχε και μια πρόταση στο κείμενό της, μια συγκεκριμένη πρόταση, γιατί ο λόγος για τον οποίο επισκεφτήκαμε τη Σικελία ήταν να παρατηρήσουμε το φαινόμενο της παρανομετανάστευσης, της υποδομές υποδοχής, αλλά και να προτείνουμε ένα συγκεκριμένο project, ένα αξιόπιστο project το οποίο θα αξιολογήσει το Κοινοβούλιο. Φοβούμε ότι αυτά τα πρακτικά, το οποίο καταγράφει τον υπερπληθισμό σε ένα κέντρο υποδοχής που περιείχε μόνο 240 ε, κλίνες και πολύ περισσότερα άτομα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εξαιρετικές υποδοχές υποδοχής, ε, εξαιρετικό προσωπικό ε, και στον Ερυθρό Σταυρό και στις άλλες αρχές της νήσου ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης του του πρόσφυγα. Είναι αληθές και ήταν σκόπιμη αυτή η αναφορά. Αλλά η Λαμπετούσα σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει να έχει ένα πληθυσμό μεταναστών που ξεπερνά τους ε, ντόπιου κατοίκους. Θα έπρεπε λοιπόν ε, να γίνει αναφορά και σε αυτό το περίεργο φαινόμενο. Ναι, είχαμε επαφέ και εμεί μη κυβερνή οργανώσει. Βεβαίω καταγράψαμε και αφιστάμενε απόψει και μεταξύ του πολύ σημαντικέ. Όμω θέλω να σα πω ότι η Λαμπετούζα είναι ένα κέντρο υποδοχή και περίθαλψη και 48 ώρε και μετά τα άτομα μεταφέρονται αλλού. Και η Λαμπετούσα είναι στο κέντρο της ε, Μεσογείου και γίνεται, αν θέλετε, στόχος ε, για πάρα πολλούς ε, μετανάστες δυστυχώς αυτό δεν ελήφθη ουσιαστικά υπόψη στα πρακτικά σας. Έπειτα, πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία με τέτοιες χώρες. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί όλο το βάρος να πέφτει στους ώμους της Ιταλίας. Μέσω των διμερών συμφωνιών, συμφωνιών που θα πρέπει να μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη αλληλεγγύη, θα πρέπει όμως να έχουμε και την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε ευρωπαϊκές συμφωνίες. Από εκεί και πέρα, κλείνοντας να πω ότι είχαμε μια εξαιρετική εμπειρία, τη ζήσαμε με όλους τους συναδέλφους, με την Γραμματεία και τους συμβούλους, όμως αυτές οι επισκέψεις θα πρέπει να οδηγούν σε ένα project, σε μια πρόταση. Ξεκινάμε από μια εξαιρετική εμπειρία που μας επέτρεψε να γνωρίσουμε πόσο καλά λειτουργούν οι άνθρωποι στην ε, επίγουσα κατάσταση υποδοχή και περίθαλψη και το πώς βοηθούν αυτούς τους μετανάστες στις πρώτες ώρες που φτάνουν στο νησί. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει πιο συγκεκριμένα να κάνουμε προτάσεις. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Μπορσελίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα περιοριστικό να μιλούμε για αποστολή στη Λαμπετούσα. Η Λαμπετούσα ήταν η αρχική επιλογή που τελικά περιόριζε την αποστολή μόνο στη Λαμπετούσα. Όμως η Λαμπετούσα είναι ουσιαστικά ένα έρημος, κατελημένος τόπος, όχι μόνο από μετανάστες. Ήταν πολύ σημαντικό να έρθουμε σε επαφή με τους ντόπιου και με τις μη κοινωνικέ οργανώσεις που ήταν οι πρωταγωνιστές στα γεγονότα που είχαν γίνει νωρίτερα όταν δηλαδή να πετούσε ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γιατί ήταν η επιλογή αυτών των δυστυχών ανθρώπων και πολλές φορές ήταν ε, ένα σφάλμα που τους οδήγησε σε αυτό το νησί και πολλές φορές μετανάστες ξεπερνούσαν τον αριθμό του ντόπιου πληθυσμού και οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση της τραγικής επίγουσα κατάστασης που τελικά αντιμετωπίστηκε και επιλύθηκε εντό εισαγωγικών αν θέλετε με αυτό τον ε, απαράδεκτο τρόπο. Με τον εκτοπισμό ουσιαστικά των μεταναστών σε άλλους προορισμούς με απαράδεκτο τρόπο. Αυτό όμως που κατ' είναι το πλέον σημαντικό και μπορούμε να κάνουμε είναι να πάψει να θεωρείται α, η Λαμπετούσα ως μη ασφαλής προορισμός. Είναι ένα στίγμα που πρέπει να εξαλειφθεί. Αυτή η έννοια, αυτό το στίγμα του μη ασφαλούς προορισμού είχε πολύ αρνητικές συνέπειες καθώς ε, Πρόσφατα προσπάθησε να προσελιμενιστεί ένα σκάφος ε, στο νησί και τελικά δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους σε κάθε περίπτωση. Εμείς παρατηρήσαμε ότι στο κέντρο υποδοχής πέρα από ένα κεντρικό στάν το οποίο είχε γίνει και μια πυρκαγιά, δεν υπήρχε τίποτα και δεν μπορούσαν πραγματικά να υποδεχθούν ανθρώπους. Επίσης και στις άλλες πόλεις Σικελίας που επισκεφτήκαμε και είδαμε τα κέντρα υποδοχής, πολλές συχνά οι συνθήκες υποδοχής ε, των μεταναστών είναι απαράδεκτες ε, και αυτό οφείλεται σε λυπή προσοχή. Η βασική, το βασικό πρόβλημα είναι τη στιγμή της υποδοχής. Και εκεί αρχίζουν ε, οι αντιπαλότητες και οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες. Όμως στο τέλος επισκεφτήκαμε και ένα κέντρο υποδοχής που ήταν εξαιρετικό. Όμως το πρόβλημα είναι η όλη καθυστέρηση της διαδικασίας που υπάρχει μετά. Ευχαριστώ η κυρία Φατζάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η αποστολή αυτή στην Σικελία, τη Λαμπεντούσα Θα ήθελα να ευχαριστώ τη συνάδελφο γιατί ηγήθηκε της ε, αποστολής μας ε, με μεγάλη επιτυχία. Εγώ θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ σε ε, κάποια αρνητικά στοιχεία, κάποιες αρνητικές εμπειρίες. Το νησί αυτό της Λαμπεντούσα έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο για τους πρόσφυγε, για του ετούντες άσυλο καλύτερο. Αυτή ο ίδιο ο ορισμό αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί πρόκειται για έναν, ορισμό, για έναν προορισμό για όλου εκείνου που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μία λύση. Πρέπει το νησί αυτό να είναι πιο ανοιχτό, να υποδέχεται εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη κατάσταση, που έχουν κινδυνεύσει να χάσουν τη ζωή του. Γιατί πρόκειται για ανθρώπου οι οποίοι ουσιαστικά πιέζονται να προχωρήσουν, να πάνε αλλού. Δεν του αφήνουν μια βραδιά να περάσουν στο νησί. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ιταλικό, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να επιδείξουν προ την ελληνική. Η δική μου εμπειρία ήταν αρνητική. Ήμουν παρούσα όταν ένας κρατούμενος στο χώρο υποδοχής εγκαταλείφθηκε σε, σε κατάσταση αντίστοιχη με αυτή που ήταν κάποιες ε, μέρες, ε, μήνες πριν. 60 σκάφη που είχαν καταλήξει στο νησί ε, εξαφανίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές μόλις πριν φτάσουμε εμείς για να μην δούμε τι συμβαίνει και φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί η πραγματικότητα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Κάποια χρήματα υπάρχουν, ναι, αλλά πολλές φορές οι υπεύθυνοι μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, και εκπρόσωποι ε, ενώσεων προσφύγων και του τον άσκηση λένε ότι δεν είναι γνωστό από τα κονδύλια που διατίθενται πόσα πάνε στην κυβέρνηση της Ιταλίας και πόσα τελικά φτάνουν στους ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Ε, δεν έχουν πρόσβαση σε εφημερίδες κρατούμενοι εκεί στο ίντερνετ, στην, ε, στις εξελίξεις στον κόσμο. Δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον κόσμο όσο μένουν στα κέντρα αυτά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πολύ πιο προσεκτικά πώς δαπανώνται τα χρήματα αυτά. Ε, κάποια θετικά που θα μπορούσα να αναφέρω, ιστορίες επιτυχίες, επιτυχίες όπως τα έλεγα, ήταν η παρουσία γιατρών εθελοντών που έρχονταν να στηρίξουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ε, πρόσφυγες, στους στο άσυλο, ε, στον ελεύθερο τους χρόνο. Συνταξιούχοι γιατροί ακόμη έρχονται και θυσιάζουν το χρόνο τους για τους ανθρώπους αυτούς πάρα πολλοί νέοι συνταξιούχοι γιατροί που βρίσκονται στην ε, Λαμπεντούσα και νομίζω ότι αυτήν, ε, αυτού του τύπου την καλή πρακτική θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Όλα αυτά καλά λοιπόν, όλα θα πρέπει να λάβουμε σαφείς απαντήσεις από τις αρχές της χώρας. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, η ώρα όμως είναι 11 πλέον, πρέπει να προχωρήσουμε το, παρα... το το μέγιστο παρακαλώ, δύο λεπτά ο καθένας, γιατί ξέρετε στις 12 και 30 αρχίζει η συνεδρία των συντονιστών και πολύ σημαντικά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε θα μας απασχολήσουν εκεί. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Παπα-Νικολάου να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν και εγώ ένας από εκείνους που ε, συμμετείχα στην αποστολή στη Λαμπεντούζα και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Βίξτρομ που ηγήθηκε της αποστολής και τη γραμματεία και όλους όσους ήμασταν μαζί και τους συναδέλφους από την Ιταλία, που εκεί είναι η κυκλογική τους περιφέρεια. Ε, ήταν ένα πολύ έντονο πρόγραμμα με διαρκή συναντήσεις και ε, πολύ σημαντική εμπειρία νομίζω για όλους μας. Ε, προσθέτοντας σε όσα ανέφεραν οι συνάδελφοι, να περιγράψω και εγώ την εμπειρία μου και τη συζήτηση που είχα με επικόους τρίτων ε, χωρών στα κέντρα που επισκεφτήκαμε που και εγώ προσπάθησα έτσι άμεσα με την επαφή μαζί τους να εξάγω συμπεράσματα. Ε, νομίζω ότι είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ για μια ακόμη φορά να τονίσουμε την ανάγκη που υπάρχει για την επίδειξη πραγματικής αλληλεγγύης στην Ιταλία αλλά και σε όλες τις χώρες που βρίσκονται ε, στα σύνορα της Ευρώπης και δέχονται έντονες μεταναστευτικές πιέσεις. Η Ιταλία τον προηγούμενο χρόνο δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις. Πράγματι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, όμως ε, σε ό,τι τουλάχιστον εγώ μπόρεσα να αντιληφθώ, διέκρινα και επαγγελματισμό, διέκρινα σοβαρή προσπάθεια, είδα σοβαρές δομές να δημιουργούνται και να εξελίσσονται ε, και αυτές είναι προσπάθειες οι οποίες πρέπει να έχουν αντίκτυπο και σε εμά ό,τι αφορά τις περαιτέρω ενέργειές μας και σε αυτά που ανέφερε βεβαίως ο κύριος Γιακολίνο πώς όλη αυτή την εμπειρία θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω και αυτό είναι μια ε, υπόθεση που δεν αφορά μόνο την Ιταλία, αφορά και την Ελλάδα που έχει αντίστοιχα προβλήματα, τη Μάλτα και άλλες χώρες, την Κύπρο που αντιμετωπίζουν τέτοιες πιέσεις. Ε, και πάλι θέλω να ευχαριστήσω. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα ακόμα. Τα πρακτικά νομίζω περιγράφουν ε, σε σημαντικό βαθμό τα όσα είδαμε εκεί και μας περιγράψανε. Οι συναντήσεις που είχαμε ήταν ε, σε βάθος, η συζήτηση και νομίζω ότι όλη αυτή η εμπειρία θα μας βοηθήσει στη συνέχεια για τις αποφάσεις που έχουμε να λάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Honorable Crocetta. Ναι, βεβαίω και εμεί να συγχαρούμε τον συναδέλφο για την δουλειά που έκανε και ιδίω τη συνάδελφο Σεσίλια, η οποία πολύ εξαιρετικά επέλυσε και κάποια διπλωματικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια τη αποστολή. Να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτή της επίσκεψη. σκεφτόμουν συνεχώς μία μόνο λέξη. Μου ερχόταν μονότονα μία λέξη. Αυτή η λέξη που φώναζαν ε, οι νέοι μετανάστες στην ε, Λαμπετούσα. Λιμπερτέ, λιμπερτέ, λιμπερτέ φώναζαν. Ελευθερία, ελευθερία, Ιταλία, Ιταλία, ελευθερία, ελευθερία. Μια λέξη λοιπόν που ερχόταν και παρερχόταν μονότονα στο μυαλό μου καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του ε, μεγάλου ταξιδιού. Ακόμα και εκεί που οι συνθήκες υποδοχές ε, ε, ήταν καλές, όπου οι συνθήκες υγιεινής ήταν καλές. Όταν κανείς φτάνει μέσα στη νύχτα μετά από πολύ δύσκολες συνθήκες ταξιδιού με ανθρώπους που δίπλα του που έχουν χάσει τη ζωή τους και έρχονται και αντιμετωπίσουν μια κατάσταση εκατανόητη, μια πολιτική εκατανόητη. Μια χώρα 60 εκατομμυρίων πολιτών. Τρίτη ευρωπαϊκή οικονομική δύναμη. Οχδοη οικονομική δύναμη στον κόσμο. 20.000 μετανάστες από την Ισία άσκησαν τόσο μεγάλη πίεση σε αυτή τη χώρα. Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα να βοηθήσουμε την Ισία με την Επανάσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα το συζητούσα το θέμα με τον ε, ε, η υφυπουργό τη την για αυτό και επεσήμανε ακριβώς αυτό το πράγμα ότι η Ευρώπη ε, επέδειξε μια μεγάλη αναισθησία σε όλο το φαινόμενο ε, και δεν υπήρξε ουσιαστικά μια παρέμβαση ανθρωπιστικού χαρακτήρα κάτι άλλο. Μήπως είναι καιρός πια να αρχίσουμε να επανεξετάζουμε το σύστημα θεωρήσεων σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία. Δηλαδή αναφέρομαι στις ε, χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολιτική προσέγγιση. Είναι παράλογο να έχουμε το ίδιο σύστημα θεωρήσεων για όλες τις τρίτες χώρες, δηλαδή με τις χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές σχέσεις, κάνουμε εισαγωγές, εξαγωγές, ε, μα τι καλά οι εμπορικές σχέσεις, αλλά τους ίδιους τους ανθρώπους τους θέλουμε γιατί φοράνε τσαντόρ, γιατί είναι μουσουλμάνοι, γιατί έρχονται από το Ισλάμ κτλ. Και τέλος. Και σε ανθρωπιστικό επίπεδο κάποια πράγματα ήταν απαράδεικτα. Όταν είδαμε το κέντρο Κάρα στο Τράπανη, εκεί είδαμε ανθρώπους ε, που έπρεπε να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου δεν είχαν πόρτες ε, ε, στις τουαλέτες. Δεν υπήρχε ζεστό νερό στο ντους, δεν υπήρχε θέρμανση. Απαράδεκτο σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Προσπάθησα να το θέσω το θέμα στον ομάρχη στο, του Τράπανη και χαίρομαι γιατί οι συνάδελφοι της αντιπροσωπείες και η ε, Σεσίλια που έθεσαν αυτό το θέμα στην Ομαρχία Τράπανη γιατί καταφέραμε να επιλύσουμε εν μέρει το ζήτημα. Πάντως θέλω να πω ότι αν δεν κάνουμε μια γενικότερη σκέψη και ε, δεν μας οδηγήσει αυτό σε επανεξέταση του συστήματος θεωρήσεων για κάποιες χώρες, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε στην Επιτροπή μας ε, με αυτό το θέμα α, οπωσδήποτε. Κύριος Μπλόμς. Διερωτώ με Πώς έγινε η επιλογή των μελών που συμμετέσχουν σε αυτή την αντιπροσωπεία. Απεστάλλει αντιπροσ... Ε, επιστολή πρόσκλησης σε όλες τις πολιτικές ομάδες αλλά και στους μη ε, εγγεγραμμένους. Γιατί εγώ δεν έλαβα καμία τέτοια ενημέρωση. Βέβαια κάποιες ε, συνεδριάσεις επιτροπής τις έχω χάσει και ίσως από εκεί να χάθηκε και η σχετική ενημέρωση. Ε, σας ε, επισημαίνω ότι οι μη εγγεγραμμένοι ενδέχεται να είχαν κάποιες παρατηρήσεις να κάνουν, ε, ίσως όχι απαραίτητα αρεστές σε όλους, αλλά πάντως δεν θα ήταν κακό να έχουν συμμετάσχει και κάποια τους μη εγγεγραμμένους. Ερωτώ λοιπόν, δεδομένου ότι άκουσα ότι είναι για κάποια τινήση μεταξύ αυτών των προσφύγων, από πού φεύγουν αυτοί οι Τινήσοι, από τι καθεστώς φεύγουν. Το καθεστώς, το νέο αυτό δημοκρατικό καθεστώς τους φάνηκε υπερβολικά δημοκρατικό και γι' αυτό δεν τους άρεσε η Τινησία και φύγανε και πήγαν στη Λαμπεντούζα. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ακούσουμε τώρα τη Σικελία. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι οι επισκέψεις στη Σικελία και τη Λεμπεντούζα ορίζονται ε, τα μέλη δηλαδή της αντιπροσωπείας ορίζονται από τους συντονιστές όπως γίνεται συνήθως. Έτσι έγινε και συγκεκριμένη περίπτωση. Για να δούμε λοιπόν πάλι τη Σεσίλια και τη Σικελία. Ευχαριστώ, λέει και Κιλία. Και ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Ε, λυπάμαι που έφυγε ο κύριος Γιακολίνο. Γιατί ζητούσε να κάνω μια ουσιαστική πρόταση. Εγώ ενήργησα εξ αντιπροσωπείας και με βάση τα συμπεφωνημένα. Συναντήθηκα με τις ε, Ιταλικές Αρχές, τους παρουσίασα μία επιστολή, τις παρουσίασα και περιμένουμε ε, απάντηση σε αυτή την ε, επίσημη επιστολή, η οποία μόλις τη λάβουμε θα σας τη μοιράσουμε. Δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι άλλο στην ομάδα. Όπως είδατε, οι εικόνες ήταν τόσο καταιγιστικές που θα τις θυμόμαστε ιστοδυναικές. Αυτό που είδα ήταν απαράδεκτο και σε καμία περίπτωση δεν αρμόσει στην Ευρώπη του 21ου αιώνα να αντιμετωπίζονται άνθρωποι όπως είδαμε να αντιμετωπίζονται. Και όλα αυτά τα δείτε στα πρακτικά. Ε, όταν ο κ. Γιακολίνο διαβάσει και τη μετάφραση στα Ιταλικά, νομίζω ότι θα συμφωνήσει με τα όσα λέει το κείμενο. Δεν θα πω και τίποτα άλλο. Θέλω απλώς ξανά να σας ευχαριστήσω για όλα. Ήταν δύσκολες στιγμές, αλλά και ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε τα, τους φραγμούς των πολιτικών οικογενειών μας, των εθνικοτήτων μας, ε, ήρθαμε κοντά χάρη σε αυτή την αποστολή και σα ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε να εκπροσωπήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προεδρέψω τις αντιπροσωπίες. Ε, μπορώ να το ξανασυζητήσω αυτό το θέμα και άλλα θέματα μαζί σας, ε, τη μετανάστευση, το άσυλο κτλ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Ε, σας ευχαριστώ για τις αρχές που προτάσετε αρχές των, της, ε, της Επιτροπής μας και που δείχνεται στους ανθρώπους που χτυπάνε την πόρτα μας ποιες είναι. Πάμε στο επόμενο σημείο. Αφορά ένα σημαντικό θέμα που έχει αντιμετωπίσει εδώ και καιρό η Επιτροπή μας. Αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 539 του 2001 περί καταλόγου τρίτων χωρών, υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών, υπήκοοι των οποίων απαπαλλάσσονται από την υποχρέωση. Ο κ. Μέρα uh, παρουσίασε το σχέδιο έκθεση στις 29 Νοεμβρίου. Ε, εν συνεχεία ακόλουθησαν κάποιες τροπολογίες, 41 για την ακρίβεια, που αφορούν τις διατάξεις, τις ασφαλιστικές δικλίδες για, τα, για τις θεωρήσεις, γρήγορη αναστολή της εξαίρεσης από την υποχρέωση θεωρήσεων. Θα μας, πει όλα, θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Δίας Δεμέρα και συνεχεία την επόμενη μισή ώρα θα συζητήσουμε το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου ευχαριστώντα του εκλεκτού συναδέλφου Επιτροπή ΛΥΠΕ, του εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του ε, Συμβουλίου για την καλή τους ε, διάθεση και στάση για την επίλυση κάποιων ζητημάτων ε, που αφορούν αυτό το ψήφισμα μας σχολείο. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Θα επιθυμούσα να υπάρχει δυνατότητα να ακουστεί δύο φορές η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, να πάρει το λόγο η Επιτροπή μετά τη δική μου τοποθέτηση και μια δεύτερη φορά αφού το ακουστούν οι συνάδελφοι. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που συζητούμε αυτή την πρώτη τροποποίηση του κανονισμού 539 και μπαίνουμε στη συζήτηση των τροπολογιών 13-54 και να πω κάτι πρακτικό. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η Τατιάνα τρεις ε, τροπολογίες για τους πράσινους, οι, οι σοσιαλιστές 14, δύο η κυρία Μπόθκουρ και πέντε η κυρία Κίνγκ. Τώρα την κυρία Βερκιά είχαμε έξι τροπολογίες όπως και τρεις του κυρίου Τρενταφυλλίδη από την ΚΟΕ. Για την κυρία Ματιέ, μία τροπολογία. Ο κύριος Βέμπερ, τρεις. Για το ΕΛΚ. Βέβερ Η κυρία Βέμπερ και ο Φιλελεύθερος, δύο τροπολογίες. Ο κύριος Κύρκοφ των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, μία τροπολογία. Και τέλος, που είναι και το πλέον ουσιώδες ζήτημα, μία τροπολογία παρουσιάστηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες εκτός του ΕΛΚ για την ενίσχυση του μηχανισμού αμοιβαιότητας, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό τον μηχανισμό. Αναφέρομαι στην τροπολογία παριθμών 28, που θα πρέπει να γίνεται κείμενο μιας πιο νυφάλιας, πιστεύω, διαπραγμάτευσης, διότι, κύριε Πρόεδρε, έχουμε να κάνουμε με μια νομοθετική έκθεση και θα πρέπει να τύχει αντίστοιχη προσέγγιση. Πρέπει ω τροπολογήσω να πω στου αδελφού ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να συζητήσω αυτή την τροπολογία στα πλαίσια τη ομάδα μου. Θέλω να ακούσω τη θέση τη ομάδα μου και να δω να έχω τη στήριξη τη ομάδα μου. Οπότε η τοποθέτηση που θα κάνω σήμερα είναι καθαρά προκαταρκτική. Τώρα για την ουσία του θέματο. Θα θυμάστε Γενικά θα πω ότι αυτή η πρώτη τροποποίηση του κανονισμού αφορά με το περιθώριο κάποιων άλλων ζητημάτων, αλλά είναι προτεραιότητας. Αναφέρομαι στην ρήτρα διασφάλισης και το μηχανισμό αμοιβαιότητας. Εργαλεία ε, με έντονο πολιτικό χαρακτήρα και πολύ σημαντικές συνέπειες, ιδιαίτερα ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον απότερο στόχο που θέλουν να επιτύχουν οι πιο πολλοί άνθρωποι που επέβαλαν τροπολογίες ό,τι αφορά τη ρήτρα διασφάλισης. με τη θέση των συναδέλφων υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αλλάξει το όνομα, να μιλήσουμε για μηχανισμό αναστολής ή να διαγραφεί και γενικότερα ο όρος και το ένα και το άλλο εγώ μπορώ να το δεχτώ. Αλλά ήμουνα εγώ αυτός ε, ε, που το είχα πει ευθύς εξ αρχής. Ό,τι αφορά την ε, σχετική τροπολογία για αυτό το μηχανισμό, πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσο αναγκαίο να έχουμε αριθμητικά στοιχεία ή ποσοστά, ως καταλητικό παράγοντα για τη διαδικασία αξιολόγησης που θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα ώστε να καθορίζουμε κατά πόσον οι συνθήκες που καταγγέλνει κάτω κράτος μέλος είναι αρκετά σημαντικές ώστε να ανασταλεί το καθεστώς απαλλαγής αποθορήσεις. Οπότε, λέω ότι πρέπει να πούμε ότι θα κινητοποιείται αυτός ο μηχανισμός αξιολόγησης, αυτή τη στιγμή αγγίζουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων, όπως αναφέρονται στην παραμετανάστες, το άσυλο, ετούτες ε, ε, επανεισδοχής που έχουν ε, απορριφθεί ασύλου. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τη γραμμή της Τάνι Αφάγιορ και αυτό που λέει το Συμβούλιο. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να προέχει είναι να, προ να μπορούμε να παρατηρούμε σημαντική αύξηση των πρακτικών συνθήκων που αντιμετωπίζει το εν λόγω κρατός Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αμοιβαιότητας, επιμένω, θα πρέπει να ενισχυθεί το κείμενο καθεστώς, γιατί πέρα και παρά από αυτό που είπε η Κομισιόν με την περίπτωση του Καναδά, είναι πράγματι αληθές ότι αυτό το κοινό σύστημα θεωρήσεως που είναι πάρα πολύ ισχυρό. Ε, και αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση αυτού του μηχανισμού και συμμεριζόμενη την θέση όλων των πολιτικών ομάδων, όπως καταδείχθηκε με την παρουσίαση κοινή τροπολογίας, την υπαριθμόν 28 δηλαδή, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τώρα, εδώ, σε αυτή τη διαδικασία ή και διμερώς αν θέλετε, ε, τις πτυχές αυτής της Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει χρόνο για να διαπραγματεύεται με τρίτη χώρα, η οποία θα ξαναεπιβάλλει την υποχρέωση θεωρήσεων. Η προθεσμία των 90 ημερών από τη δημοσίευση της τροποποίησης σε 45, που είναι η πρόταση στην τροπολογία 28, την κοινή τροπολογία, θεωρώ ότι δίνει πολύ μικρό περιθώριο λιγμών για διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ λίγο το περιθώριο των 45 ημερών και ιδίω αν λάβουμε υπόψη και τις πολιτικές σχέσεις και άλλου χαρακτήρα που διακυβεύονται με τρίτη χώρα. Για αυτό το λόγο, στην πρώτη μου έκθεση, στο πρωταρχικό κείμενο, προτείνω να χρησιμοποιήσουμε το μέγιστο αριθμό των 90 ημερών και μόνο στην περίπτωση όπου οι συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν ότι δεν πηγαίνουμε σε μια συμφωνία, να ξεκινάει η διαδικασία τη συναπόφαση για την ε, προσωρινή επαναφορά τη απέτηση θεωρήσεων ε, στην τρίτη χώρα ε, με την οποία συζητούμε. Επίση, η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να παρατείνεται αυτή η διαδικασία θα μπορούσε και πάλι να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ή, αν θέλετε, για να συνεχίσει να πιέζει, με άλλα λόγια. Στην περίπτωση που η τρίτη χώρα επανεξετάζει τη θέση της, κάθε αυτή την περίοδο, τότε ε, αρκεί για να αποσυρθεί η πρόταση αυτή. Έπειτα, θέλουμε μία διευκρίνηση, Τάνια παρακαλώ, μία διευκρίνηση σχετικά με τον μηχανισμό που προβλέπετε στην τροπολογία σας, όπου θα μπορεί να επιβληθεί μετά την προθεσμία των 90 ημερών, ώστε να επαναφέρει την, την αυτόματη υποχρέωση θεώρηση. Επίσημα αυτό, αυτόματη επαναφορά θεωρήσεων. Και θα ήταν αναγκαίο να κατανοήσουμε και να μας ε, πείσετε αν θέλετε για το κατά πόσο είναι βιώσιμη νομικά αυτή η λύση. Εγώ δεν έχω ουσιαστική ένσταση, αλλά νομικά δεν ξέρω κατά πόσο στέκει. Οπότε, ε, επαναλαμβάνω αυτή την προσωπική μου θέση και θέλω να δω αν θα έχω την υποστήριξη της πολιτικής μου ομάδας. Ε, κύριε Πρόεδρε, Σας ε, ευχαριστώ επίσης για τη διευκρίνηση που κάνατε στο ερώτημά μου στον Δανό Υπουργό. Γιατί είναι ένα ερώτημα στον Δανό Υπουργό ε, γιατί κατανοώ ότι η απάντησή του ήταν η σιωπή. Δεν απάντησε καθόλου. Και αυτό μας δίνει μια εικόνα, Τάνια και αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο περίπλοκο πολιτικά είναι αυτό το ζήτημα που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχει μεγάλη ικανότητα ρητορική, ε, αλλά ελάχιστη έως μηδαμινή ικανότητα να λαμβάνονται αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ΑΦΕΤ, όπου ζητά να λαμβάνονται υπόψη εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης κατά τη στιγμή επανεξέταση, επαναφοράς ε, ε, της επιβολής των θεωρήσεων. Θα ήθελα να πω ότι οι σχετικές ε, γνωμοδοτήσεις της Frontex, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου και της Europol να έρθουν να προσταθούν σε αυτά και η σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων. Ευχαριστώ εν προκειμένου τον κύριο Κόβατσεφ. Στις διαπραγματεύσεις τώρα που είχαμε με την ε, προσωπικούς του Συμβουλίου θέλω να πω ότι ήταν εξαιρετική η πρόθεση του Συμβουλίου για την αύξηση, αν θέλετε, του, της συμμετοχής, της ενεργού συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις όλες τις διαπραγματεύσεις. Πάντω, ο, ο μηχανισμός θα πρέπει να κινείται με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα. Το κατανοούμε αυτό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να λαμβάνει αποφάσει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα. Συμφωνούμε και δημόμαστε προ αυτήν την κατεύθυνση. Στην δεύτερο γύρο τη τοποθέτησής μου, κύριε Πρόεδρε, θα πω συγκεκριμένα και με σαφήνεια ποια είναι η αρχική μου θέση για την κάθε μία από τις τροπολογίες. Επιμένω όμως, ο τροπολογία 28 που είναι αν θέλετε και το ψητό, να το πω έτσι λαϊκά, θα πρέπει να τύχει μιας νυφάλιας διαπραγμάτευσης και να δούμε κατά πόσο νομικά στέκει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον Δία, Θεμέρα για την παρουσίαση της έκθεσης και για το τοποθετική και τις 42 τροπολογίες. Και όπως και εσείς προτείνατε, ναι, καταγράψαμε και εμείς πόσο πολιτικά ευαίσθητο είναι το ζήτημα. Κατανοούμε ότι θέλετε και εσείς τη στήριξη πρώτα απ' όλα πολιτικής ομάδας για αυτές τις τροπολογίες. Και επίσης κατανοούμε ότι είναι καλό να υπάρχει μια γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας ε, του Κοινοβουλίου για το κατά πόσο είναι νομικά αποδεκτές κάποιες τροπολογίες. Το δεχόμαστε. Να ακούσουμε τώρα τι έχει να πει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιάν Τεκόιστερ. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά και πάλι να πω ότι έχω ένα μακροσκελή κατάλογο αγοριτών, αλλά σας το λέω της εξ αρχής, μόνο δύο λεπτά. Διότι στις 12 η ώρα έχουμε την παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου, τον κυρίου Βίσερ. Για να μπορέσουμε λοιπόν να διαχειριστούμε καλά το χρόνο, παρακαλώ πρώτα απ' όλα και την Επιτροπή να κρατήσει το χρόνο, αλλά και δύο λεπτά για το κάθε συνάδελφο. Και μετά θα κλείσει ο κύριος Διεθνέμερα, ο κύριος Ντεκόιστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα Ήθελα να εστιαστώ στα δύο ζητήματα που έθεσε ο, που έθεσε ο εισηγητής, καταρχάς τους μηχανισμούς αμοιβαιότητας και δεύτερον τον μηχανισμό άρσης. Ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ στον μηχανισμό αμοιβαιότητα, στο άρθρο 28, τη δυνατότητα δηλαδή να εξασφαλίζονται συνενέσεις μεταξύ των διαφορών ομάδων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε κάποιε αμφιβολίε ω προ την ε, νομική ορθότητα τη πρόταση αυτή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανονικά, δηλαδή, ένα κράτο το οποίο καθίσατε διαπιστώνει ότι είναι θύμα ε, μη εφαρμογή αρχή τη αμοιβαιότητα πρέπει να κοινοποίηση στην Επιτροπή και βέβαια μπορούμε να ενημερώσουμε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δημοσιεύεται λοιπόν αυτή η κοινοποίηση και στη συνέχεια με 45 μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για να θέσει πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις ε, μία αμοιβαιότητας. Και λέμε στο άρθρο 28 ότι θα διαπιστώσει την επανόρθωση Τη κατάσταση στην θεώρηση διαβατηρίων. Δηλαδή δεν μα δίνει κανένα περιθώριο διακριτικό αυτό το άρθρο. Ε, δεν θα θέλαμε όμω του αυτοματισμού, γιατί μάλλον δυσκολεύουν το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ίδιο ο εισηγητή είπε ότι θα πρέπει η, εξωτερική, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να έχει περιθώριο να επαληθεύσει το μηχανισμό αυτό, όπως προτείνει άλλωστε και η Επιτροπή ΑΦΕΤ και η περίπτωση της μη αμοιβαιότητας και η πιθανότητα αποκατάστασης αμοιβαιότητας ε, θα πρέπει να ε, κρίνεται με βάση και πτυχές εξωτερικών σχέσεων και άλλα ζητήματα. Άρα, ο τόσο σαφής ε, αυτοματισμός που ορίζεται στο άρθρο 28 για την Επιτροπή δεν είναι αποδεκτός. Επιπλέον, ο αυτοματισμός που προβλέπεται μου γεννά και άλλη αμφιβολία και προβληματισμό. Αναφέρεται δηλαδή συγκεκριμένα στο κείμενο ότι μετά την υποβολή τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την ακμή των 45 ημερών δηλαδή, θεωρείται ότι εάν δεν έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συναπόφασης που να πάβει τον μηχανισμό αυτόν, θεωρείται ότι έχει ήδη υλοποιηθεί. Αυτή η γιοτίνα δηλαδή, η λεμιτόμος, μερικές φορές όντως μπορεί να τεθεί από το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ε, κίνηση για ε, λόγους εξωτερικών σχέσεων. Ερωτώ όμως τότε, τι εξυπηρετεί ο αυτοματισμός στην αμοιβαιότητα εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν έχουν επαρκή πλειοψηφία, μάλλον έχουν επαρκή πλειοψηφία για να ρίξουν την κοιλιοτίνα. Τι θα πώς μπορούμε να πιέσουμε μια τρίτη χώρα Αφού δεν υιοθετείται η πρόταση, δεν μπορούμε να έχουμε πια περιθώριο να πιέσουμε, δεν έχουμε μοχλοποίηση για τη τρίτη χώρα. Άρα θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε, πιστεύω, για έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό αμοιβαιότητα. Αλλά δεν είμαστε καθόλου πεπισμένοι ότι ο αυτοματοποιημένο αυτό μηχανισμό εξασφαλίζει ψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τη ρήτρα διασφάλιση, που μετατρέπεται τώρα σε μηχανισμό άρση διακοπή, και δεν έχουμε αντίρρηση ω προ την αλλαγή ορολογία, Πιστεύω ότι τα κριτήρια της θέσης σε εκείνης είναι το κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή, Συμβούλιο, Επιτροπή, Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι θα πρέπει για εξαιρετικέ περιστάσει να προβλέπεται ένα τέτοιο μηχανισμό ε, άρση τη λειτουργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω γνωρίζετε, προτείνει διαδικασία ε, επιτροπολογία και έχει διορίσει μαθηματικά, αριθμητικά κριτήρια δηλαδή για την θέση εκείνη τη διαδικασία και βέβαια πρέπει να γίνει αξιολόγηση τη κατάσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη όλων των σχετικών περιστάσεων και ιδιαίτερω και ζητημάτων ε, ε, μελημάτων εξωτερικών σχέσεων. Το Συμβούλιο από την άλλη πλευρά εγκαταλείπει αυτά τα επακριβή και μετρήσιμα κριτήρια και τα αντικαθιστά από μια αναφορά σε μια ε, άξαφνη ή ξαφνική και σημαντική αύξηση. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε να ρωτήσουμε το Κοινοβούλιο τι γνώμη έχει για τα κριτήρια αυτά. Στην προηγούμενη μα συζήτηση είχαν επευθυνθεί επικρίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η προσέγγιση που ακολουθεί είναι μαθηματικού χαρακτήρα. Θα ήθελα όμω να υπογραμμίσω πω πιστεύουμε ότι αυστηρός προσδιορισμένα κριτήρια, συγκεκριμένα κριτήρια, είναι ακριβώ αυτά τα οποία αποτελούνται για να τίθεται σε κίνηση ο μηχανισμός. Και τότε δεν θα υπάρχει πια αυτοματοποιημένο σύστημα. Θα πρέπει με μία πολιτική απόφαση να προτείνει ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άρση του καθεστώτος θεωρούς διαβατηρίων. Αλλά όχι μόνο αυστηρά και μόνο μαθηματικά κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Σα ακούσουμε τώρα του συναδέλφου. Σα υπενθυμίζω ότι έχουμε μόνο δύο λεπτά στη θέση μα. Έκαστο. Το Συμβούλιο έχει εκπρόσωπο. Στο κοινοβούλιο, στην αίθουσά μας είσαστε εδώ παρόντες, παρούσα. Μέρχαμ, παρακαλώ, από το Συμβούλιο. Θέλετε να μιλήσετε πριν αρχίσουμε τη συζήτηση. Δεν θέλετε. Ορίστε, δεν θέλει κιόλα. Ευχαριστώ. Βεβαίω, Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια που μας κάνατε για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από τον εισηγητή και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και για την ε, θαυμάσια συνάντηση που είχαμε χθες όπου είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Ε, άκουσα ότι ο Δανός υπουργό δεν απάντησε πραγματικά στο ερώτημα, αλλά το ερώτημα είναι πολύ λεπτό. Και δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει το Συμβούλιο τη θέση του για το αν θα υπάρξει αυτοματοποίηση ή όχι. Είναι ένα σημαντικό θέμα επί Προεδρίας και ελπίζω οι Υπουργοί να καταφέρουν να ανοίξουν τη διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο και όταν γίνει αυτό να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Σε ομάδα εργασίας πάντως θέλουμε πολύ να προχωρήσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ενδεχομένως ελπίζω να τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Λοιπόν, δύο λεφτά στον καθένα τώρα. Ο κύριος Μπουσουτήλ, πρώτος και καλύτερος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Ντία Στεμέρα, όχι μόνο για την παρουσίαση, αλλά και για την προσέγγιση με την οποία προσέγγισε αυτό το θέμα. Ανοιχτή προσέγγιση. Θα ήθελα να μιλήσω για το μηχανισμό αναστολή καταρχήν. Ένα μηχανισμό αναστολή και η ρήτρα διαφύλαξη, πέστε την όπω θέλετε, χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι εκ των όνου κάνευ. Εγώ είμαι υπέρ τη αυτοματοποίηση, δεν είμαι πεπισμένο από τα επιχείρηματα τη Κομισιόν για την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχει για την πρωτοβουλία και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό το σημείο να το κάνουμε ε, θεσμική διελκυστήντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, ρεαλιστικοί στην προσέγγισή μας. Τελικά ένα συμπέρασμα βγαίνει όταν βλέπουμε τι γίνεται. Σήμερα δεν έχουμε ένα κοινό σύστημα θεωρήσεων. Όταν μία ή περισσότερες χώρες στυλιτεύονται ή αφήνονται στο περιθώριο από τρίτες χώρες ε, στα πλαίσια του συστήματος ε, θεωρήσεων, μένουν μόνες τους στο κρύο. Και μέχρι στιγμής η Κομισιόν δεν τις βοήθησε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά τη χώρα μου, που είναι η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από 8 χρόνια, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήσ, βγάλαμε την υποχρέωση θεωρήσεων για τους ε, Βραζιλιάνους. Ήταν απαραίτητο με βάση τον κώδικα θεωρήσεων. Το κάναμε λοιπόν. Μετά από 8 χρόνια, οι πολίτες μας, μαζί με τους πολίτες ακόμα τριών ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται ακόμα θεώρηση για να πάνε στη Βραζιλία, για να ταξιδέψουν στη Βραζιλία και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι αποτυχία του συστήματος ε, αμοιβαιότητας. Επί 8 χρόνια. Και οι πολίτες μας έχουν βαρεθεί. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε κοινό σύστημα θεωρήσεων αν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα, ένα τρόπο υπάρχει να το κάνουμε. Δηλαδή, όταν μια τρίτη χώρα συνεχίζει να εργή, χωρίς κανένα λόγο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα αυτόματο σύστημα το οποίο αναστέλει τα ωφέλη, θα πρέπει αμέσως να τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Τατζάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντία Στεμέρα, ευχαριστώ τους Σκιώδης, ευχαριστώ την Δανέζικη Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι η μέχρι τούδε συνεργασία μας ήταν θαυμάσια. Θα ήθελα να τονίσω δύο θέματα μόνο, ούτως ώστε είμαι και εντός των χρονικών ορίων. Έχουμε αυτό το μηχανισμό αναστολής και τη ρήτρα προστασίας. Είναι ένας πολιτικός μηχανισμός που θα χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός τελικής καταφυγής. Είναι μια λύση κατεπίγουσα. Είμαστε σε μια παράδοξη φάση, κατάσταση. Ανοίξαμε την πόρτα σε πολλές χώρες πρόσφατα, παραδείγματος χάρη στα Δυτικά Βαλκάνια, και τώρα συζητάμε ήδη πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα μηχανισμό για να κλείσουμε αυτή την πόρτα που ανοίξαμε. Ελπίζω να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτός ο μηχανισμός. Χαίρομαι που αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν και που διαγράφουμε νούμερα, ποσοστά κτλ. Οι μαθηματικοί τύποι δεν είναι οι κατάλληλοι για να προσεγγίσουμε τις ακραίες καταστάσεις. Στη δική μου τροπολογία, ή μάλλον στις τρεις δικές μου τροπολογίες που έχω υποβάλει, ε, προτείνω να διαγραφούν αυτά τα ποσοστά. Μιλάω μόνο για κατεπίγουσες καταστάσεις, για ταχύ αύξηση των ε, ετούντων ε, άσυλο ή των προσφύγων και πρέπει να βελτιώσουμε το κείμενο εκεί που λέει ότι δεν θα πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα αναγκαστούμε να κλείσουμε την πόρτα σε όλους όσους ε, ζητούν άσυλο ή είναι πρόσφυγες και που έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Ελπίζω αυτή η κατάσταση να μην ξανασυμβεί στο μέλλον και να μην κλείσουμε την πόρτα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα στο άσυλο. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούμε σε αυτή τη διαδικασία από την αρχή στο τέλος. Βασίζομαι στην γνωμοδότηση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και νομίζω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μόλι λαμβάνει έκθεση από οποιοδήποτε κράτο ε, μέλο που ισχυρίζεται ότι έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με μια τρίτη χώρα. Μέσα σε τρει μήνε η Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογεί την σοβαρότητα τη κατάσταση και θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσα σε αυτό το διάστημα των τριών μηνών. Και συνεχεία τα, αυτά τα δύο θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο Συμβούλιο, θα πρέπει να γνωμοδοτούν με τη σειρά του μέσα σε ένα μήνα. Ε, δεν θέλουμε οι κανόνε τη επιτροπολογία να παρακάμπτονται, αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενταχθεί στην όλη διαδικασία και να συμμετάσχει. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αμοιβαιότητα, θα είναι δύσκολο το σημείο, το βλέπω στις διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνω όλες τις ανησυχίες και τις συστάσεις ε, του εισηγητή. Χρειαζόμαστε μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, αλλά ο μηχανισμός αμοιβαιότητας δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε. Και οι μικρές χώρες δεν θα πρέπει να μπαίνουν στη γωνιά να στριμώχνονται από τον Καναδά ή τι ΗΠΑ από μεγάλε χώρε, δηλαδή μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν αρκετά μέσα για να αντιδράσουν. Μιλάω για την Τσεχία, Φερρυπίν ή την Αυστρία, τέτοιε χώρε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε απειλούν την Αυστρία ότι θα την ε, βγάλει από το πρόγραμμα εξαίρεση ε, από τι θεωρήσει, αν δεν επιτρέψει η Αυστρία στι ΗΠΑ να, έχει πρόσβαση, να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Προβλέπω σκληρέ διαπραγματεύσει. Η δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2010 ε, προσκαλεί την Κομισιόν να δημιουργήσει ένα νέο μηχανισμό που θα εξασφαλίσει πλήρη αμοιβαιότητα για όλα τα κράτη-μέλη και που θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη που δεν είναι τα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούν να παραβιάζουν αυτό το μηχανισμό αμοιβαιότητας. Ε, και σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση, όλα τα κράτη-μέλη θα επαναφέρουν την υποχρέωση ε, θεωρήσεων για αυτή την τρίτη χώρα. Αυτό ε, υπάρχει στη δήλωση του Κοινοβουλίου του 2010 και νομίζω ότι αυτή η γραπτή δήλωση θα πρέπει να προταχθεί. Περιμένω, λοιπόν, σκληρές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε δελεχή συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις και όπως σας είπα ήδη, πιστεύω ότι ο μηχανισμός αναστολής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κανονικά. Το δικαίωμα στο ταξίδι είναι το δικαίωμα που πρέπει να έχει κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Ο επόμενος θα πρέπει ε, ο μηχανισμό αναστολή να είναι μηχανισμό τελευταία καταφυγή. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ακριβώ. Δεν πρέπει να παίζουμε παιχνίδια τώρα με αυτόν τον μηχανισμό. Πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά. Να σκεφτούμε τη διατύπωση ε, του μηχανισμού αυτού αναστολή. Ήδη έχω ένα πρόβλημα. Μιλάμε για μηχανισμό κατεπίγουσα ανάγκη. Α το σκεφτούμε. Α είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίση, χρειαζόμαστε ένα σαφέστατο μηχανισμό για να αποφύγουμε τις αυθαίρετε αποφάσεις. Ε, συμφωνώ κύριε Μπουσούτη, δεν έχουμε κοινό σύστημα θεωρήσεων. Θα, πρέπει θα έπρεπε να έχουμε. Είμαι έτοιμη να αρχίσουμε ή μάλλον να συνεχίσουμε τις συζητήσει. για την τροπολογία 28. Αν δημιουργεί νομικά προβλήματα, ας το συζητήσουμε ξανά. Συμφωνώ απόλυτα. Και ας ζητήσουμε τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας, όπως είπαν κι άλλοι. Καταλαβαίνω γιατί τη ζητάτε. Πάντως, εγώ θέλω να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός, ο οποίος να είναι όμως σαφέστατος, εναντιέστατος. Η κυρία Φαγιάν είπε ότι δεν χρειαζόμαστε ποσοστά και νούμερα. Συμφωνώ. Αλλά θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, αν ξεφορτώθουμε τα νούμερα οι μαθηματικοί τύποι είναι αόριστοι, υπάρχουν τεράστια περιθώρια ερμηνείας ε, Το βασικό είναι να μην έχουμε περιθώρια διαφορετικών ερμηνεών. Ε, κοιτάξτε την τροπολογία 33. Λέμε ότι πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα, αλλά ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα συνολικό νούμερο ε, ε, υπηκών των χωρών και να πάρουμε αποφάσεις από αυτή τη βάσεως. Επίσης, τροπολογία 35, κοιτάξτε την. Όπου εκεί είμαστε ακόμη πιο ακριβείς, έχω την αίσθηση, σε ό,τι αφορά την ρήτρα αναστολή. Όταν ειδικά υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, ε, σωματεμπορία... Έχω την εντύπωση ότι αν είμαστε πιο ακριβείς, βελτιώνουμε τα πράγματα παρότι συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοσοφία της κυρίας Φαγιάν, μήπως μερικές φορές χρειαζόμαστε κάποια όμως, κάποια λίγα αριθμητικά στοιχεία, για να μην αφήσουμε τεράστια περιθώρια ερμηνείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντίας Δεμέρα, τους Κιώδης. Ελπίζω να πετύχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα αποδεκτό, ικανοποιητικό. Άκουσα τον κύριο Ντεκώστα. Αρχίζω να κατατρώγομαι από αμφιβολίες. Τροπολογία 28, αμοιβαιότητα. Που την ε, συνυπέβαλαν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Υπάρχει, και εκεί λέμε, μας λέτε κύριε Ντεκώστα, είναι αποτελεσματικός αυτός ο μηχανισμός αυτοματοποίησης. Έχει απλώς προληπτικό χαρακτήρα. Η τρίτη χώρα δεν θα ξέρει ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει. Και θα αρχίσει να ρωτάει, πρέπει να ξεχωρίσουμε μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βάλουμε εκεί την υποχρέωση θεωρήσεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να το ξέρει ότι υπάρχει. για τη ρήτρα αναστολή. Μακάρι η νομική υπηρεσία να εγκρίνει τη θέση μας για να προχωρήσουμε. Για αυτό το μηχανισμό αναστολής υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Στην ομάδα μου προτείνουμε το 50% να, πάει, να γίνει 100%, ε, άλλοι λένε 60%, άλλοι μιλάνε για ουσιαστική αύξηση. Ε, ποια είναι η ουσία, να υπάρξει μια ουσιαστική, όταν υπάρχει ουσιαστική αύξηση. Να δούμε τι γίνεται. Μια και ξέρω από μαθηματικά. Η αριθμητική είναι πολύ μικρό τμήμα των μαθηματικών. Ελπίζω να βρούμε ένα καλό μαθηματικό τύπο, εν πάση περιπτώσει, για αυτά τα ποσοστά. Κυρία Ρόιτοβα. Eh, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ όλους τους συζητητές, όλους τους συναδέλφους που αγωνίζονται, που προσπαθούν να δημιουργήσουμε εν τέλει ένα ενιαίο σύστημα θεωρήσεων, κάτι που μας λείπει Ελπίζω να με ακούτε καλά. Τα κράτη-μέλη έχουν δεμένα τα χέρια. Κατά τη διάρκεια διμερών επαφών, κάνουν ό,τι μπορούν ενώ πιέζονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς παρακολουθεί αυτές τις διαπραγματεύσεις και δεν πιέζει καθόλου τις τρίτες χώρες να επαναξιολογήσουν την αρχική τους θέση και να λάβουν υπόψη κάποια νέα δεδομένα που θα μπορούσαν να απαιτούν την επανεισαγωγή της υποχρέωσης θεωρήσεων ή αντίστροφα. Είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα και πρέπει να έχει μια στεναρή στάση. Η εθνική μας αντιπροσωπεία υποστηρίζει την ε, τροπολογία 21 και σε ό,τι αφορά τον, την αυτόματη εφαρμογή της αμοιβαιότητας, ε, τροπολογία 28. Μέχρι το 2001 υπήρχε αυτή η αυτόματη εφαρμογή. Και το χρησιμο... τη χρησιμοποίησαμε στο πακέτο των 6 προτάσεων. Δεν πρέπει να, να φοβόμαστε αυτό το μηχανισμό, γιατί δεν είναι καινούριο. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα, αλλά μια κοινή πολιτική θεωρήσεων με αυτό τον αυτόματο χαρακτήρα θα πρέπει να έχει ε, ανασταλτικό χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να βάζουμε την υποχρέωση θεωρήσεων όπως να είναι, ας πούμε. Θα πρέπει να έχουμε στεναρούς λόγους. Για... Η... η έκθεση έχει κάποιες σωστές παραδοχές. Ε, κοινή πολιτική, γιατί κοινή είναι μια άλλη ιστορία. Είναι βασικό στοιχείο για να ελέγξουμε την ε, λαθρομετανάστευση. Πολλέ τρίτε χώρε, πολλοί υπήκοοι, έχουν υποφεληθεί από την εξαίρεση τη θεωρήσεων και ζητούν διεθνή προστασία ε, χωρί κανένα λόγο ή λίγου λόγου. Φυσικά ασχολείται με το μηχανισμό ε, αναστολή και λέει ότι ο μηχανισμό θα πρέπει να ξεκινήσει να δρομολογήσει μια διαδικασία αξιολόγηση. και εν συνεχεία θα πρέπει να υπάρξει δράση μόνο όταν υπάρχει ουσιαστική αύξηση στη λαθρομετανάστευση. Γιατί αυτή η καθυστέρηση, για να μπουν πάρα πολλοί δηλαδή οι λαθρομετανάστε. Η έκθεση λέει ότι θα ήταν αντιφατικό να θεωρήσουμε τις θεωρήσεις ε, ως αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης. Διαφωνώ δεν είναι προβληματική και ούτε ακριβό αυτό το εργαλείο, ούτε χρονοβόρο, μπορούν να εκδοθούν πάρα πολύ γρήγορα, ηλεκτρονικά κτλ. Ε, όταν κάποιο μπαίνει σε μια χώρα ε, και όταν βγαίνει, απλώ το καταγράφουν. Ε, εγώ όταν πηγαίνω στην Αυστραλία στην οικογένειά μου το καλοκαίρι, ε, μου εκδίδουν ε, μια θεώρηση. Αν παραμείνω παράνομα στο τέλος της διαμονής, τότε αυτό θα το καταλάβουν οι αρχές και είναι πολύ σωστό να το καταλάβουν και να το εντοπίσουν. Θα πρέπει να υπάρχουν θεωρήσει για όλε τι χώρες, από τις οποίες υπάρχει ουσιαστική τάση, λόγο ο πληθυσμό τους να έρχεται εδώ πέρα στην Ευρώπη. Ε, επίσης, ε, η αμοιβαιότητα ε, νομίζω ότι γίνεται από ε, τράγος. Αποκλείεται ε, να μεταναστεύσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι μαζικά προς φτωχές τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ακούσατε όλα αυτά τα σχόλια του Ευρωβουλευτέ. Η Κομισιόν, η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει πριν δώσω ξανά το λόγο για τα τελικά σχόλια στον κύριο Ντία Δεμέρα. ευχαριστώ. Για το μηχανισμό αναστολής. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για τον ορισμό των κριτηρίων. Λοιπόν, ε, όταν μιλούμε για επίγουσα κατάσταση, δεν πιστεύω ότι αρκεί ούτε να μιλάμε για μια κάποια αύξηση της ε, πίεσης. Ταυτόχρονα είπατε ότι πρέπει να, ο μηχανισμός αναστολής να είναι η ίστατη λύση και ελπίζουμε να χρησιμοποιηθεί ποτέ. Για αυτό το τελευταίο συμφωνούμε κι εμείς. Όμως φοβούμεθα ότι όσο πιο ασαφές και θολό είναι το κριτήριο εκείνης του μηχανισμού, τότε πιο ψηλός είναι ο κίνδυνος α, στο μέλλον, το μέλλον να τον κινήσει αυτό το μηχανισμό. Να το έχετε και αυτό υπόψη κατά τη διάρκεια των συζητήσεών σας. Τώρα, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μηχανισμό αναστολής από την ε, αρχή των συζητήσεων για αυτή την πρόταση εμείς είπαμε ότι έχουμε δεσμευτεί πολιτικά να έχουμε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Βεβαίως, αυτό θα πρέπει να γίνει θεσμικά α, με καλό και ορθό τρόπο. Άρα λοιπόν να τηρούμε τις αρχές τους, και τους κανόνες επιτροπολογίας ώστε να βρούμε την πλέον κατάλληλη λύση και αυτή συνεργασία. Και τέλος ένα πολύ σοβαρό και δύσκολο ζήτημα που είναι ο μηχανισμός αμεβαιότητας. Ποιο συνάδελφό σα μίλησε για το καθιστό 2001 που δεν περιείχε τέτοια ρήτρα, ναι πράγματι. Όμως ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Μόνο ένα κράτος μέλος κίνησε το μηχανισμό αυτό πριν το νέο μηχανισμό αμοιβαιότητας που δεν είναι αυτόματος τέθη σε ισχύ. Κανένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποίησε τον αυτόματο μηχανισμό και άρα ποτέ αυτό δεν επηρέασε τρίτες χώρες από επιβάλλουν θεωρήσεις. Για τη συνολική αποτελεσματικότητα του κείμενου συστήματος, πρόεδρε, μου επιτρέπετε, δεν θέλω τώρα να φανώ εχθρικός, ε, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς στην Κομισιόν είμαστε πεπισμένοι ότι ο μηχανισμός αυτός ήταν επαρκής για τις πάνω από 100 με βιότητας κυρίως με τις ΗΠΑ και τον Καναδά είχαμε κάποια προβλήματα, κάποια κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ακόμα το πρόβλημα και έπειτα υπάρχει και το θέμα της Βραζιλίας που έθεσε κάποιος συναδελφό σας, πράγματι, αλλά να σε επενθυμίσω ότι έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσεις για ε, ένα αμοιβαίο σύστημα απαλλαγή αποθόρη με τη Βραζιλία, που αυτή τη στιγμή είναι κατά τη διαδικασία κύρωση από το Βραζιλιανό Κοινοβούλιο. Έχουμε έρθει σε επαφή με τις ε, αρχές Βραζιλίας για να πιέσουν και να προχωρήσουν την κατάσταση. Όμως, ξέρετε, το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο έχει την απόλυτη κυριαρχία και αυτονομία και αποφασίζει τους χρόνους κατά τους οποίους θα κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, ασκούμε πίεση, αλλά μέσα σε κάποια όρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ε, συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να καταστήσουμε το μηχανισμό πιο αποτελεσματικό. Αλλά για να καταλήξουμε σε μια πλήρω κοινή πολιτική, κοιτάξτε, ακόμα και η τροπολογία 28 δεν μπορεί να εγγυηθεί ε, μια ε, κοινή πολιτική. Διότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την αναστολή του αυτόματο χαρακτήρα. Δεν μπορείτε να εγγυηθείτε τη στάση της χώρας. Αν τρίτη χώρα δηλαδή επαναφέρει προσωρινά την αναστολή των θεωρήσεων, Πώς μπορούμε λοιπόν να κινηθούμε κοινά. Πρόεδρος, θέλει το Συμβούλιο να τοποθετηθεί. Αν όχι, θα δώσω το λόγο για τελικό σχόλιο. Στον... Θέλει το, το Συμβούλιο, παρακαλώ, εντάχει. Eh, Σας ευχαριστώ. Άκουσα τα σχόλια βεβαίως για την ε, έκθεση, τις τροπολογίες και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε πιστεύω σε εις βάθεως διαπραγματεύσεις. Όταν μιλάμε για αμοιβαιότητα, δεν χωρεί αμφιβολία, ότι τα κράτη-μέλη στηρίζουν το Κοινοβούλιο στα θέματα της αμοιβαιότητας στη θεώρηση των Πιστεύω ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να το εμπλέξουμε στη δικασία αυτή να δυνατόν πιο νωρί. Και βεβαίω να προσδιορίσουμε και το ρόλο των θεσμικών οργάνων, ε, ώστε να έχει το καθένα τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται, να αντιδρά όταν πρέπει ε, ταχαίω ε, έναντι των τρίτων χωρών και να κοιτάξουμε να προσδιορίσουμε τι βασικέ αρχέ και αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τι βασικέ αρχέ, δηλαδή την αμοιβαιότητα προς το παρόν δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειε. Έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε συνεδρία τη ομάδα εργασία ε, αργότερα που θα το, που, όπου θα το συζητήσουμε. Ο κύριο Διάστε Μεϊρά για να καταλήξουμε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο που μου δώσατε, το οποίο διαχειρίζεστε πολύ καλά παρά τι θα πρέπει να πω πρώτα πρώτα ότι λυπούμε για μια παράληψη. Θα πρέπει να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Πολωνική Προεδρία για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να προωθήσει αυτή την πρόταση. Ο κύριος Κούστερ και η Επιτροπή Εν Γέννη. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, ακρίβεια και αμεσότητα στα λεγόμενά σας. Και μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευτυχέ αυτό το γεγονός, άσχετα αν συμφωνώ ή όχι με όλα όσα είπατε. Ναι, σας ευχαριστώ για τις προθέσεις σας ε, να δώσετε μεγαλύτερο ρόλο σε ειδικές επιτροπολογίες στο Κοινοβούλιο. Τα ακόμη προσοχή, ακόμη προσοχή και αυτά που είπε η Ιδανική Προεδρία. Η Ιδανική Προεδρία είπε τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν το Κοινοβούλιο. Για να το δούμε και αυτό στην πράξη. Πάντως μας ικανοποιεί και μόνο αυτή σας η Ευχαριστώ τον Σάιμον, την Τάνια για τα σχόλια που ήδη τα γνώριζα. Για την κυρία Έρνστ, τροπολογία 33 και 35. Θέλετε ποσοστά και θέλετε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όταν μιλούμε για δικηματικές πράξεις. Τατιάνα, ο μηχανισμός με μία διάσταση πρόληψης, είπατε. Ούτε εσείς θέλετε αριθμητικά στοιχεία. Και τη μαθηματικός δεν θέλετε αριθμητικά στοιχεία. Θέλετε να μιλούμε για σημαντική αύξηση. Έπειτα, ευχαριστώ την κυρία Ροϊτόβα του ΕΛΚ που ε, προσυπέγραψε και αυτή την τροπολογία 28 παρά τα αυτά ε, και αυτή συμφωνεί για την διάσταση πρόληψη που πρέπει να έχει μηχανισμό. Ο κ. Μπρόγκ είπε ότι η αμοιβαιότητα δεν είναι σημαντική, κατά τη γνώμη του. Τώρα, συγκεκριμένα πράγματα μπορώ να πω, αλλά προκαταρτικά. Σε σχέση με τις τροπολογίες που υπευλήθησαν για το ΕΛΚ, ο κύριος Ματιέ υπέβαλε μια τροπολογία, μπορώ να δεχτώ, ο κύριος Βέμπερ, τρεις τροπολογίες, δεκτές και αυτέ. Ο κύριο, η κυρία Βέμπερ των Φιλελευθέρων δύο τροπολογίες υπέβαλε και οι δύο δεκτές. Ο κύριος Κύρικοφ των Στηρητικών μία τροπολογία δεκτή της ε, Δημοτικής Αριστεράς Κυριάκος και Κορνέλια τρεις τροπολογίες που προς το παρόν απορρίπτονται. Και πάλι, Κορνέλια και Κριστίνα, έξι τροπολογίες που τις δέχομαι. Δέχομαι τέσσερις. Απορρίπτω μία και την άλλη μπορούμε να την πραγματευτούμε. Θα έχω επαφές με όλους τους συναδέλφους για τις περαιτέρω διευκρινήσεις. Σε ό,τι αφορά τους δημοκράτες, η Τάνια υπέβαλε τέσσερις τροπολογίες, δέχομαι δύο και τις άλλες δύο θα τις δούμε, τις δεν Μεταξύ αυτών είναι και η περίφημη 28. Ο κύριος Εντιέ. Μία τροπολογία την οποία δέχομαι. Κύριο Ποθκούρ, δύο τροπολογίες. Μπορούμε να τις συζητήσουμε και τις δύο ότι παραπέμπουν στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ έχω την ε, τροπολογία 7, μπορείτε να τη δείτε, θα το συζητήσουμε πάντως. Κυρία Κίνια, την Αντιπρόεδρο, πέντε τροπολογίες, δέχομαι τις τέσσερις, απορρίπτω τη μία. Για τους πράσινους, να πω στην Τατιάνα που υπέβαλε τρεις τροπολογίες, εξαιρετική δουλειά έκανε, δέχομαι τις δύο, απορρίπτω πέντε, αλλά μπορώ να διαπραγματευτώ άλλε έξι. Αυτά συνοπτικά, Πρόεδρε. Πρέπει να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο τη συζήτηση για την τροπολογία 28 και την τροπολογία 10 που συνδέονται μεταξύ. Δηλαδή η 10 είναι η δική μου και η 28 είναι η ομαδική τροπολογία από τις πολιτικές ομάδες. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Διεθεμ Λασμέρα. Όχι μόνο γιατί με την παρουσίαση και τα συμπεράσματά σας συμβάλλατε στην καλή διαχείριση του χρόνου, αλλά γιατί λάβατε υπόψη και όλα τα σχόλια και της Προεδρίας Συμβουλίου και της Κομισιόν και μας δείξετε και τη διάθεσή σας έναντι των τροπολογιών. Ποιες δέχεστε, ποιες απορρίπτετε, ποιες θα συζητήσετε, ώστε οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που ήταν παρόντας εδώ γνωρίζουν ακριβώς τη θέση του εισηγητή για να ορίσουμε καλύτερα τη διαδικασία από εδώ και πέρα. Βλέπω ότι ο κύριο Δεθμέρ θέλει ένα τελικό σχόλιο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε για την κατανόηση, θα είμαι πολύ σύντομο. Ξέχασα κάτι που μου έδωσε ο Αλεξάνδρα Άλβαρο, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Σκόπιμο θα ήταν να το λάβει υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και η νομική υπηρεσία Λέει ο Αλεξάνδρου ότι υπάρχει προηγούμενο σε ό,τι αφορά τον αυτόματο χαρακτήρα του μηχανισμού και μου αναφέρει την, το πρόσφατα ε, εγκεκριμένο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, το λεγόμενο six-pack. Η 1173 του 11, 1174 του 11 και 1175 ε, του 2011 με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2011 είναι αποφάσεις του, του Συμβουλίου συγγνώμη, που ε, περιέχουν τον ίδιο αυτόματο χαρακτήρα. Αυτό μου λέει ο κύριος Άλβαρο. Εγώ το πιστεύω και παρακαλώ να καταγραφεί και να ληφθεί υπόψη. Και από τη δική μας νομική υπηρεσία στη γνωμοδότηση της και να το λάβει υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, συμφωνώ, λέει ο Πρόεδρος. Καταγράφουμε αυτό το τελευταίο σας σχόλιο, κύριε Τίας Δεμέρα, και είναι σαφές ότι πλέον ζητούμε γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, ώστε να διασκεδαστούν οι αμφιβολίες ερωτηματικά που ακούστηκαν για τις ρήτρε διασφάλισης και αμοιβαιότητας. Καλώς? Ωραία. Για το επόμενο μισάωρο περνούμε να συζητήσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης πριν κάνουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Βίσερ, τον κύριο Ρόμπερτ Βίσερ, τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου, της ΕΑΣΟ, με άλλα λόγια, να σας καλωσορίσουμε κύριε Βίσερ. Θα σας δώσουμε το λόγο να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα εργασίας 2012 του Γραφείου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Mr. Chairman, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά που με προσκαλείτε στις αρχές του χρόνου, του 2012. Παρακαλώ, ησυχία λέει ο πρόεδρος. κύριος Φίσερ έχει ήδη ανάψει το μικρόφωνο του, σας υπενθυμίζω. Παρακαλώ. Όποιος σκοπεύει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει ησύχω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις αρχές του νέου έτους, λοιπόν, του 2012, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Θα υπενθυμίσω ότι Αρχίσαμε να εργαζόμαστε το 2011, άρα το 2012 θα είναι το δεύτερο πλήρε έτο. Το 2010 ξεκινήσαμε, το 2012 λοιπόν θα είναι το δεύτερο πλήρε έτο λειτουργία τη ε, υπηρεσία μα. Ξεκινήσαμε βέβαια προσπαθώντα να ε, χτίσουμε από το μηδέν την υπηρεσία. Ξεκινήσαμε διάφορα συγκεκριμένα θέματα. Ιδιαίτερο με την προσπάθεια να στηρίξουμε την Ελλάδα στι ιδιαίτερε δυσκολίε που αντιμετώπιζε σχέση με το άσυλο. Θα δείτε βέβαια ότι έχουμε ένα ευρύτατο πεδίο καθηκόντων από τον κανονισμό μας που θα μας απασχολήσουν και φέτος και θα ήθελα ξεκινώντας ε, να αναφέρω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να περιγράψω καλύτερα τη δουλειά μας. Η υπηρεσία στόχο έχει να στηρίξει το κοινό σύστημα ασύλου σύγκληση στην πράξη, καθημερινή πρακτική και στήριξη στην ε, καθημερινή προσπάθεια των κρατών μελών μέσα στο κοινό σύστημα ασύλου. Έτσι λοιπόν, η υπηρεσία μας εστιάζεται σε τρία-τέσσερα κύρια στοιχεία. Στήριξη στη βάση στο σημείο δηλαδή όπου διαπιστώνεται ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη σύγκληση, κατάρτιση, εκπαίδευση. Με ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης που έχουμε εισαγάγει καταρχάς, ε, που να εξασφαλίζει ότι θα ε, ε, έχουν όλοι την ίδια αντίληψη, την ίδια κατάρτιση, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε την κοινή κατάρτιση για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε σύγκληση των δράσεων, του τρόπου εργασίας καλύτερα. Δεύτερον, θέλουμε να έχουμε ε, αξιόπιστες πληροφορίες για τη διαδικασία του ασύλου μέχρι την λήψη της αποφάσεως που ε, διεξάγεται σε μία χώρα, ανάλογα με την χώρα προελεύσεως. Εφόσον λοιπόν ε, οι πληροφορίες αυτές είναι αξιόπιστες, αντικειμενικές, αμερόληπτες, μπορούμε πιστεύω να συμβάλλουμε και ίσως είναι καλύτερη αυτή η συμβολή στη διαδικασία ασύλου που θα διεξαχθεί με, που θα μπορέσει να έχει πολύ ψηλή ποιότητα. Επίσης, θέλουμε ένα σύστημα συναγερμού προειδοποίησης. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι σε διάφορα κέντρα συζητήσεων αναπτύσσεται διάλογος για ένα σύστημα εγκαίρης προειδοποίησης, όπως ονομάζεται στο δικό μας κανονισμό Ήδη προβλέπεται ένα τέτοιο σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση, ένα σύστημα συνογερμού, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή εφέτος και θα δίνει πληροφορίες για την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη και κατά τρόπο συγκρίσιμο που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Και ως προς τις ε, προς τις ικανότητες, το δυναμικό δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο έχουν τα κράτη-μέλη χτίσει το σύστημά τους, αλλά και ως προς το εξωτερικό, ε, το τι μπορούμε να προβλέψουμε ή να αναλύσουμε σαν εξελίξεις. Βέβαια δεν, δεν ε, ισχυρίζομαι ότι μπορούμε να προβλέπουμε το μέλλον, αλλά μπορούμε ενδεχομένω να αναλύουμε εγκαίρω δεδομένα ώστε να βλέπουμε από πού μπορεί να έρχονται κάποιε ροέ και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα προπαρασκευαστικά, ελπίζω τουλάχιστον εγκαίρω, μέτρα. Ακόμη ένα άλλο τμήμα, αλλά εξίσου σημαντικό, η αρχή της αμοιβαιότητας, της αμοιβαιότητας ε, που σημαίνει ότι πρέπει να οργανώσουμε δράσεις αμοιβαιότητας, αλλά και ιδιαίτερες δράσεις, όπως συνέβη με την Ελλάδα, επί παραδείγματι. Μέχρι τώρα και ε, συζητήσεις που συνεχίζονται ακόμη με ένα άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να του προσφέρουμε έκτακτη ε, στήριξη με βάση την αμοιβαιότητα. Την ελεγγύη καλύτερα. Και άλλα στοιχεία του προγράμματος εργασίας μας είναι η ιδιαίτερη μένυμνα για τους ε, ασυνόδευτους ανήλικους. Η εξωτερική δράση θέλεις, χρειάστηκα να λάβω απόφαση και πρέπει να πω ότι δεν μου ήταν καθόλου ευχάριστο γιατί αποτελεί σημαντικό τμήμα του φακέλου για την ε, μετανάστευση. Αναγκάστηκα λοιπόν να αποφασίσω να αφήσω το θέμα αυτό κατά μέρος για αυτή τη χρονιά γιατί ίσως να αποδειχθεί, αποδεικνύεται καλύτερα ε, απαραίτητο κάτι τέτοιο λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων, των δημοσιονομικών περικοπών που υπέστη η υπηρεσία μου. Ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια να είναι διαφορετική η κατάσταση και επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστώ θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξη και την τροπολογία του. Εν πάση περιπτώσει εκφράστηκε ιδιαίτερη υποστήριξη προς την ε, υπηρεσία μας από πλευρά του Κοινοβουλίου και στη δημοσιονομικά. Επίσης, Πρόεδρε, Στην ακροασή ε, μου, 9 του 2010, είχα υποσχεθεί στο Κοινοβούλιο ότι θα οργανώσω ένα συμβουλευτικό φόρουμ με την κοινωνία των πολιτών ε, μέσα στον πρώτο χρόνο της ανάληψης των καθηκόντων μου. Στις 15 Δεκεμβρίου πέρυσι έγινε ε, το πρώτο αυτό συμβουλευτικό φόρουμ στην Βαλέτα της Μάλτας όπου με χαρά είδα εκπροσώπηση και της Επιτροπής ε, των Πολιτικών Ελευθεριών με την κυρία Τζιν Λάμπερτς. Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος ήταν μια καλή αρχή. Διάλογος με την ε, κοινωνία των πολιτών δεν σημαίνει μια σειρά από συνεδριάσεις μόνο και πάντως όχι μια μόνο συνεδρίαση, μια μόνο εκδήλωση, αλλά πάντως ε, θα αποτελέσει μια αλληλουχία, μια σειρά, μια ολόκληρη οργάνωση και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα θετικό απολογισμό από αυτή την ε, ε, εκδήλωση. Στον απολογισμό εκεί επίση, Πρόεδρε, θα ήθελα να σημειώσω ότι το να χτίσει μια υπηρεσία από το μηδέν δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Πολλέ ήταν οι δυσκολίε που αντιμετωπίσαμε. Αλλά τώρα πια έχουμε μια υπηρεσία με, ε, τα, ε, γραφεία στη Μάλτα, με ένα προσωπικό 35 ατόμων στη Μάλτα την ίδια και με 10 περίπου άτομα προσωπικό στο γραφείο πασάρ των Βρυξελών. Πάμε καλά δηλαδή. Έχουμε ένα προσωρινό κτίριο προς το παρόν στη Μάλτα. Ελπίζω ότι μέχρι τα μέσα του έτους θα έχουμε το δικό μας τελικό κτίριο και έτσι ε, θα μπορέσουμε, ελπίζω να έχουμε και προσωπικό μέχρι 60 ατόμων να αυξήσουμε το προσωπικό μας. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσει η συζήτηση. Ας ξεκινήσει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κ. Τζούλι Ντιμπλάζη. Δεν θέλετε. Όχι. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε. Από την 1η Φεβρουαρίου του, 2000, του πέρυσι έχετε αναλάβει το αξιωμά σας. Ε, σας έχουμε αφήσει έτσι μια περίοδο χάριτος, αλλά τελείωσε τώρα και ελπίζουμε ότι το 2012 θα, μας, θα υπάρξουν αποτελέσματα. Ε, το Κοινοβούλιο ήταν υπέρ της δημιουργίας αυτής της υπηρεσίας, αυτού του οργανισμού και τώρα ανυπομονούμε για να μας παρουσιάσετε αποτελέσματα σε ένα τομέα που μας ενδιαφέρει τα μάλλα. Να κάνω τρεις ερωτήσεις. Ε, σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Δανό Υπουργό της ε, Προεδρίας να μας λέει ότι αύριο θα θέσει το θέμα του μηχανισμού πραγματικής αλληλεγγύης ε, επιτάπητος στο τραπέζι του Συμβουλίου επιτάπητο ε, στο Συμβούλιο Τζάι. Υπάρχει η πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν για την ε, αλληλεγγύη. Ε, πέστε μας, το γραφείο σας, το ΕΑΣΟ, ε, έχει εμπλακεί στη δημιουργία αυτού του, πραγμα... του... μηχανισμού αλληλεγγύης για το πρόγραμμα επανεκατάστασης ε, για τη Μάλτα. Η, η ΕΑΣΟ θα έχει ένα ρόλο στην επέκταση αυτού του προγράμματος ούτως ώστε όχι απλώς να γίνει μόνιμο, αλλά να αφορά όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία θα μπορούν ε, δυνητικά να υποφεληθούν από αυτό. Ασχολείστε ήδη με το πρόγραμμα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ήταν πολύ επιτυχημένο. Τρίτον, η Άσο μελετά ή συνεισφέρει στην ε, συνεχιζόμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Ο κανονισμός του Δουβλίνου μπορεί να έχει κολλήσει, αλλά όσο είναι κολλημένος, το δικαστήριο της, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εκδίδει τις αποφάσεις του και τώρα θα παίρνουμε αποφάσεις που θα λένε ότι έτσι όπως έχει ο κανονισμός του Δουβλίνου, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί μπορεί να παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα. Συμμετέχει η Άσο σε αυτή τη συζήτηση για το του Δουβλίνου, που είναι σημαντικός ε, και εσωτερικό, στοιχείο, αν θέλετε, του πακέτου για το άσυλο, αυτός ο κανονισμός. Λόπες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίσερ για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Πραγματικά περιμέναμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τις εμπειρίες σας μετά από ένα έτος σε αυτή τη θέση. Πρέπει όμως να πω ότι οι γενικές γραμμές του προγράμματος εργασίας σας, όπως μας εκθέσατε, είναι ανεπαρκείς. Διότι δεν μπήκατε στην ουσία, θα χρειαζόμαστε μια εις βάθος ε, παρουσίαση του έργου του γραφείου σας για να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα ύπαρξη του γραφείου. Χρειαζόμαστε, αν θέλετε, περισσότερες λεπτομέρειες και πιο πολλές πληροφορίες για τις οποίες λαμβάνετε βάση των οποίων εργάζεστε. Δηλαδή, τι πληροφορίες παίρνετε από τις εθνικές κυβερνήσεις, πόσα είναι τα κέντρα υποδοχής που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα στις χώρες του Νότου. Ρωτώ. Ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο. Μπορεί να μην έχουμε ένα επίσημο σύστημα συλλογή δεδομένων για αυτό το θέμα, αλλά πόσα τέτοια κέντρα υποδοχή έχουμε, πόσο είναι ο χρόνο παραμονή σε αυτά τα κέντρα κράτηση, πόσο είναι ο χρόνο αναμονή για να λάβουν μια απάντηση στην αίτησή του πόσους αιτούντες άσυλο έχουμε βάσει το κανονισμού του Δουβλίνου ε, και πώς επιλύεται το θέμα, το είτε μέσω καθεστώς ε, επικουρικής προστασίας και πόσοι τη χάνουν επιστροφής. Αυτά είναι ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε όταν μιλούμε για άσυλο. Αν δεν μπαίνετε σε τέτοιες λεπτομέρειες εμείς ως ευρωβουλευτές, ε, ε, κινούμεθα στα τυφλά. Ο λόγος δημιουργίας ε, του ΕΑΣΟ ήταν αυτός, για να αποκτήσουμε μια τέτοια ακριβή εικόνα. Τουλάχιστον ρωτώ, θα ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να σας δίνουν τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνήσεων, να σας δίνουν αυτά τα στοιχεία. Έχουμε την αίσθηση ότι οι αιτούντες άσυλο βρίσκονται σε μια κατάσταση χειρότερη και από τον τελευταίο εγκληματία. Δεν έχουν δικονομικά δικαιώματα. Ζουν σε ε, ικτρές συνθήκες. Έχουν χειρότερη μεταχείριση και από τους τελευταίους ε, φερόμενους εγκληματίες της Ένωσης. Ρωτώ λοιπόν, έχετε ουσιαστικές πληροφορίες ή πώς μπορείτε να καταλήξετε στο να λαμβάνετε ουσιαστικές ε, και βάσιμες ε, πληροφορίες για την κατάσταση ασύλου, για την συνεργασία ή μάλλον για την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Θα θέλαμε και πολλές λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια πειραματικά προγράμματα που αφορούν αυτή την αλληλεγγύη. Ρωτώ, Μιλούμε ουσιαστικά για μια αλληλεγγύη που ε, δόθηκε για περίπου 300 ε, ετούτε άσυλο. Μα απ' την άλλη έχουμε πλημμυρίδα, έχουμε χιλιάδες ετούτε άσυλο στα κέντρα υποδοχής. Τι γίνεται με αυτούς. Δηλαδή αυτά τα πειραματικά προγράμματα, να αφορούν κάποιες λίγες εκατοντάδες άτομα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πλημμυρίδα των ατόμων που περιμένουν. Αυτά γνωρίζουμε και αυτό μα λένε και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και όσο κρατάει αυτή η κατάσταση, αυτό είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Παπα-Νικολάου. Uh, Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ε, είμαι Έλληνας. και ασχολούμαι εδώ, στις διαπραγματεύσεις, ε, εδώ στην Επιτροπή για τις με τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο ασύλου. Προσπαθώ να παρακολουθώ τις εξελίξεις ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαδικασία του ασύλου και τα επίπεδα προστασίας που παρέχουμε. many of our discussions... Σε πολλές από τις συζητήσεις μας με τους ενδιαφερόμενους, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με συναδέλφους, με άλλα θεσμικά όργανα. Αναφερόμαστε στην ΝΕΑΖΟ ως ένα νέο εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για να βρούμε λύσεις σε πολλά θέματα που διαπραγματευόμαστε σε πολλούς φακέλους που προσπαθούμε να προωθήσουμε. Φερρυπίν. Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό του 2. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα εργασίας ε, του 2012 ότι το προσωπικό είναι το προσωπικό υποστήριξη για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού έγκαιρη προειδοποίηση αποτελείται από ένα άτομο. Συμφωνώ ότι προσπαθούμε να στήσουμε μια υπηρεσία από το μηδέν. Έγιναν συζητήσει ε, για την ΕΑΖΟ. Σε αυτέ τι συζητήσει κάθε φορά υποστηρίζουμε την ε, ΕΑΖΟ, γιατί πιστεύουμε σε αυτήν την υπηρεσία. Οι άλλοι όμω μου λένε ότι η υπηρεσία είναι νέα, ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη, σας επισημαίνω αυτά που είπε ο κύριος Μπουσουτήλ και, ο κύριος Λόπες Δεμέρο. Ε, η, η ΑΖΟ όντως θα πρέπει να γίνει ο, ο εμπειρογνώμονάς για τι διαδικασίε ασύλου στην Ευρώπη. Αυτό έχουμε στο μυαλό μα. Να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν εμπειρογνώμονα, μια υπηρεσία α πούμε με η δημοσύνη για να υποστηρίζει κάθε κρατό μέλο. Σε αυτή την κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή η Άζο μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του η Δήμονα. Τα οικονομικά σας, όπως είπατε, δεν είναι αυτά που έπρεπε να είναι. Πέραν τούτου, όμως, η εντολή σας είναι η ενδεδειγμένη μπορείτε χάρη σε αυτή την εντολή να δημιουργήσετε αυτή την πραγματογνωμοσύνη και να βρείτε λύσεις στα προβλήματα της διαδικασίας ασύλου. Πες τα ελληνικά. Κυρία Αγγελίλη. Κυρία Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλωσορίζω τον κύριο Βίσερ. Τρεις ερωτήσεις. Οι πρώτες δύο έχουν γίνει από τον κύριο Μπουσουτήλ βέβαια τις ε, προσυπογράφω και εγώ. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου στη συζήτηση για το μηχανισμό για την ελληνική και την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο 2. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Ξέρουμε ότι το θέμα αυτό είναι κατεπήγον. Οι ανήλικες είναι ευάλωτα πρόσωπα πρέπει να τα προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως. Γι' αυτό η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών ζήτησε και πέτυχε από την Επιτροπή ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ένα πιλωτικό σχέδιο για αυτό το θέμα των ανηλίκων. Συχνά οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι τοπικές αρχές ασχολούνται με αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο. Και μάλιστα το κάνουν χωρί να έχουν επαρκή πόρου για να το κάνουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, αυτά τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή. Δεν πρέπει απλώ να τα υποδεχτούμε. Πρέπει να πάνε σχολείο συχνά. Πρέπει να τα υποστηρίξουν ψυχολογικά, να δουν ένα ψυχολόγο. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ σωστά. Πρέπει να υπάρχουν και ανθρώπινοι πόροι ε, πρέπει να υπάρχουν επαγγελματίε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οικονομικοί πόροι για, αυτό, για αυτή την πλαισίωση. Εσεί αναφερθήκατε έτσι σε αυτό το εμπαρόδο σε αυτό το θέμα, αλλά θέλω να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματιώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Διευθυντά. Δύο ερωτήσει από μένα. Καταρχά, την... μας μιλήσατε για την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Πετε μα περισσότερα πράγματα και για Πεςτε μας και κάτι παραπάνω για τις σχέσεις που έχετε με την ε, υπηρεσία Frontex. Ο κ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να ρωτήσω ψηφοφόρους γιατί χρειάζεται μια κοινή πολιτική ασύλου. Ίσως ο λόγος είναι να προσπαθήσουν οι κυβερνήσεις να προστατευτούν από την πίεση της κοινή νόμας του κάθε κράτους μέλους ως προς τις πιέσει αυτές του ασύλου. Έτσι λοιπόν μπορούν να να συγκαλύπτονται πίσω από την ε, πλασματική ευαισθησία και απόγνωση στην οποία περιέλχονται και να υποκρύπτονται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά όμως αυτή η υπηρεσία δεν έχει καμιά πραγματική ευθύνη, ευθύνη και χρησιμοποιώ τη λέξη εσκεμένα, δηλαδή ούτε λογοδοσία, ούτε έχει, ούτε μπορεί κανεί να την παρετήσει από τους πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κοινοβούλιο όμω έχει ευθύνε. Όμω δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα θεσμικό όργανο από όλα του πλέγματος Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια κανένα πολίτη δεν μπορεί να γνωρίζει ο κάθε ευρωβουλευτή τι πρεσβεύει και σε ποιο βαθμό. Ίσως θα πρέπει με τι επόμενε ευρωεκλογές να το θυμίσουμε. Ευχαριστώ, λίγο ο και εσεί τώρα παρακαλώ για να μα δώσετε τι απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ τις κυρίες και κυρίους βουλευτές για τις ε, παρατηρήσεις τους. Και πάνω απ' όλα που μου υπενθυμίζουν ότι τέλειωσαν οι γλύκες, τέλειωσε ο μήνας του μέλητος και πρέπει πια να προσφέρουμε, να αποδείξουμε ότι προσφέρουμε έργο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εύστοχη η παρατήρηση ότι θα πρέπει στο δεύτερο αυτό έτος η Επιτροπή, η υπηρεσία να λειτουργεί σωστά, να αποδίδει έργο και όχι να αποτελεί απλώς δαπάνη κονδυλίων. Επιτρέψτε μου τώρα από τι διάφορε ερωτήσει που ακούστηκαν να δώσω κάποιε απαντήσει, ενδεχομένω να κάνω και κάποιε πιο γενικέ παρατηρήσει. Για το αν εμπλεκόμαστε στον ε, μηχανισμό αλληλεγγύη και τη συζήτηση για το Δουβλίνο 2, η απάντηση είναι ναι. Αύριο θα είμαι στο Συμβούλιο ε, Δικαιοσύνης και Ιστορικών και θα δώσω απαντήσεις. Γενικά έχω συμμετάσχει στη συζήτηση που οδηγεί σε κάποιες προτάσεις και πιστεύω ότι η υπηρεσία μας έχει τέτοιο ρόλο να διαδραματίσει. Και με το σύστημα της προειδοποίησης, το early warning όπως ονομάζεται, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για τον κύριο Παπανικόλα. Εάν είναι σε θέση η υπηρεσία μας να διαδραματίσει το ρόλο αυτόν κάποια στιγμή. Εδώ νομίζω ότι έγκυται ακριβώς η ουσία του ζητήματος. Ως υπηρεσία με περιορισμένους πόρους και την οποία περιμένουν ε, τεράστιες προσδοκίες, βλέπω ότι είναι δύσκολο το έργο. Η εμπειρία μέχρι τώρα είναι θετική, αλλά χρειάζομαι υποστήριξη. Υποστήριξη από κάθε πλευρά. Και για να συνεχίσω με το θέμα της ενημέρωσης και της ε, αυτό είναι δυνατό, δηλαδή είναι δυνατό να θεσπιστεί ένα σύστημα ενημέρωση έγκαιρη προειδοποίηση, όπως προτείνει η κυρία Λόπε, μόνο εάν συνεργαζόμαστε, αν υπάρχει συνεργασία. Με καταπλήσει λοιπόν το γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αλφα ιστορία πίσω τη. Το θέμα του ασύλου δε και των προσφύγων, 10-15 χρόνια τουλάχιστον ιστορία. Για ορισμένε χώρε ακόμη μεγαλύτερη ιστορία και εμπειρία. Και όμω ακόμη δεν έχουμε συγκρίσιμα αξιόπιστα και ανεξάρτητα δεδομένα πληροφορίε. Φυσικά και αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να ε, αντιμετωπιστεί μέσα σε μερικέ εβδομάδε ή μήνε. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται να οργανώσουμε, να συλλέξουμε τι πληροφορίε από τα κράτη-μέλη, να τι οργανώσουμε και για την ερώτηση του κ. Πανικολάου, εάν η εντολή τη υπηρεσία μα αρκεί, θα έλεγα ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο στόχο είναι, αναφέρεται στον κανονισμό. Αναφέρεται κάποια μορφή ε, διάχυση πληροφοριών και σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση. Αλλά τυπικά δεν έχω το δυναμικό για να απαιτήσω από τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τον ένα ή τον άλλον ορισμό ή να δίνουν την τάδε ή τη δίνα πληροφορία ή τα δεδομένα. Νομίζω ότι είναι δυνατόν μέσα στην ε, δομή και με τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η υπηρεσία μας να οργανωθούμε κατά τρόπον ώστε να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή Και έτσι, εδώ και καιρό, και δεν έχω αρκετό προσωπικό, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί βέβαια ε, δικαιολογία. Θα συνεχίσουμε από τον Εύρο έχουμε ξεκινήσει, θα συνεχίσουμε να, δια, να συλλέγουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και στην ετήσια μας έκθεση θα συμπεριλάβουμε τα στοιχεία αυτά. Ελπίζω ότι έχουμε σε αρχές του, της δηλαδή Μάρτιο ή Απρίλιο, με περιεχόμενο. Φυσικά πρόκειται για μια πρώτη έκθεση και έτσι θα χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, αλλά θα περιλαμβάνει, φαντάζομαι, τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες τη θέση των, την ανεξάρτη, τις ανεξάρτητες θέσεις των εμπειρογνωμόνων που σωστά απαιτείτε και εσείς να τις περιλάβουμε. Και αυτό αφορά όχι μόνο τη Eurostat και τα κράτη-μέλη, αλλά και συγκεκριμένα τις μη κυβερνητικέ οργανώσει. Προσπαθούμε να έχουμε δηλαδή στον δυνατό στοιχεία από αυτά που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σημείο επανεγκατάστασης ε, και τη Μάλτα. Πολύ σημαντική παρατήρηση, αλλά ιδιαίτερος και λόγω της ανακοίνωσης Επιτροπής θέλεις του 2011. Ότι η επανακατάσταση θα πρέπει να προβληθεί περισσότερο στην πολιτική μας. Έχω προτείνει υποστήριξη για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας ε, επανεγκατάστασης που είναι ακόμη υπό προετοιμασία και άρα πρέπει να πω ότι προς το παρόν δεν συμμετέχω ενεργά. Αλλά θα γίνει αυτό άπαξ και ενεργοποιηθεί η δεύτερη φάση. Να εδώ τι άλλο μπορεί να έχω λησμονήσει. Ασυνόδευτη ανήλικη βεβαίως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στη διαδικασία αυτή Εμεί τρόπον την στο θέμα αυτό είμαστε η υπεργολάβη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Είναι μια ευρωπαϊκή εμβέλεια ε, δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά του ανηλίκου, ε, του αθνόδου ανηλίκου και δεν αφορά μόνο την ίδια τη δουλειά τη υπηρεσία μα. Είναι πολύ ευρύτερο, καλύπτει διάφορα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή και με τη Frontex. Πάνω σε αρκετέ διαφορετικέ δράσει στο πρόγραμμα δράση. Στηριζόμαστε σε δύο βασικά θέματα. Πρώτον, αξιολόγηση της ηλικία σε όλες τις πτυχές τη. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και γενικότερα, πέραν της ηλικία πώς αντιμετωπίζουμε πώς χειριζόμαστε το θέμα των συνόδων ηλικών, Με μεγάλη σημασία στην ηλικία και βέβαια προσπαθούμε να συλλέξουμε ευέλικτε πρακτικέ και γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ από, από και για τα κράτη-μέλη και για τι υπηρεσίες μη κυβερνητικέ οργανώσει. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει βεβαίω εμπλέκονται και σε αυτή τη διαδικασία στι συζητήσει μα για την κατάρτιση. Πρόγραμμα κατάρτισης είχε ξεκινήσει κατά πιλωτικό τρόπο στη λεγόμενη διάσκεψη GDASC Από 1η Ιανουαρίου του 2012 έχουμε αναλάβει εμεί. Αρχικά είχαν συμμετάσχει τα κράτη-μέλη. Τώρα όμω έχουμε εμεί αναλάβει το λεγόμενο EEC, δηλαδή European Asylum Curriculum, ω σχέδιο και θα αναλάβουμε το τρέξιμό του για το 27, ίσω και 28 από του χρόνου κράτη-μέλη. ώστε να αποτελέσει αυτό το κύριο βασικό πρόγραμμα κατάρτισης. Γενικά παρακολουθούμε ποια είναι τα ε, προγράμματα σπουδών, τα προγράμματα κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου για να προκύψει ένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργασία με τη Frontex βεβαίως σε πολλούς συγκεκριμένους τομείς αναφέρθηκα στους ε, ασυνόδευτους ανηλίκους γιατί η Frontex έχει ρόλο στην αναγνώριση, στον εντοπισμό στο σύν, στα σύνορα των ασυνόδευτων ανηλίκων, αξιολόγηση κινδύνου επίσης, αλλά και έγκαιρη προειδοποίηση αφού στοιχεία συλλέγει και η Frontex, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται επικάλυψη εργασία. Στην Ελλάδα Φερρυπίν συνεργαστήκαμε με το ελληνικό πρόγραμμα δράσης το οποίο αφορά και το άσυλο αλλά και τη διαχείριση των σύνορων ταυτόχρονα. Συνεργαστήκαμε με τη Frontex. Επίσης, άλλοι τομεί στους οποίους ε, κοιτάμε αν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία, ε, κατάρτιση, κατάρτιση προσωπικού από διάφορες υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις. Για δε τη λογοδοσία προσωπικός, θεωρώ τιμή μου να είμαι η πρώτη υπηρεσία υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας που έχει πιο ουσιαστικό ρόλο και κατά κάποιον τρόπο και την υποχρέωση λογοδοσία, όπου έχει κάποιο πιο ουσιαστικό ρόλο και την λογοδοσία και τον ελέγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή δουλειά για το 2012. Ευχαριστώ για όλες τις ε, παρεμβάσεις συναδέλφους. Περάσαμε για λίγα λεπτά το χρόνο μας και γι' αυτό ευχαριστούμε και τους διερμηνείς που μας έδωσαν λίγο παραπάνω χρόνο. Σας ευχαριστούμε κύριε Φίσερ και ευχόμαστε ότι καλύτερο. Ένα λεπτό μόνο διακόπτω ώστε να αποχωρήσουν όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα γιατί θα γίνει και κλεισμένο.